Good Κυρίες και κύριοι, ας αρχίσουμε με την συνεδρίασή μας. Ορισμένες ανακοινώσεις ε, καταρχήν. Αποφασίσαμε στους συντονιστές να ισχύσει η νέα διαδικασία γνωμοδοτήσεων σε σχέση με τις τροπολογίες. Πρόκειται για το πολιετές πλαίσιο των πελαγικών ειδών στην Αδριατική θάλασσα η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι ανοιχτή για τα μέλη της ΕΜΒΗ και στη συνέχεια θα υποβληθούν ε, οι τροπολογίες σε ψηφοφορία. Εκείνες που θα εγκριθούν θα υποβληθούν στην Επιτροπή Αλίας από εμένα, από την Πρόεδρο, εξ ονόματος της Επιτροπής μας και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 23η Ιουνίου στις 11, στις 11 το πρωί. Μία δεύτερη ανακοίνωση αφορά την κοινή εκδήλωση για τους στόχους, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις 7 Ιουνίου. Αποκινούμε την Επιτροπή Ανάπτυξης και οργανώνεται από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη ε, με τον υπεύθυνο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι παρόν και ο, πρόεδρος της Νορβηγίας καθώς και ο πρόεδρος Ταγιάννη στα δύο πάνελ για τους ε, βιώσιμους στόχους και θα έχουμε τέσσερις εκπροσώπους από τον ΟΗΕ. Ελπίζω να είσαστε πολύ παρόντες. Σήμερα έχετε και την έκθεση της επίσκεψης στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλ. και σήμερα έχουμε 20 γλώσσες και όπως ξέρετε η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά και αναμεταδίδεται απευθείας η συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται και τα πρακτικά μας της 13ης Μαρτίου. Σήμερα ο πρώτος μας ε, εισηγητής είναι ο κύριος Ζίγκβιτ Μουρεσάν που είναι γενικός εισηγητής για το 2018 και θα ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό και θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης στην διαδικασία προϋπολογισμού όπως έχει συντονιστεί και ο τριμερής διάλογος θα λάβει τη μορφή μιας επιστολής η ΕΜΒΗ έστειλε 40 σχέδια γνωμοδότησης για πιλωτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, η έκθεση γνωμοδότησης θα λάβει χώρα στη... θα ψηφιστεί στις 10 ε, Ιουλίου και στη συνέχεια θα εγκριθεί και από την Ολομέλεια. Δίνω το λόγο στον κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε σήμερα. Ε, σήμερα το απόγευμα ήρθα για δύο λόγους για να σας υποβάλω τις απόψεις μου για τις ε, βασικές πολιτικές ε, προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό για του χρόνου, όπως τις εγκρίναμε στις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018, το Μάρτιο, κατά την Ολομέλεια και θα ήθελα να ακούσω τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2018, έτσι ώστε να ξέρω τι είναι σημαντικό για σας και τι θα πρέπει να λάβω υπόψη. Όπως είπε και η Πρόεδρος, οι δύο προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2018 είναι η ανάπτυξη και θέσεις εργασίας καθώς και η ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό το έκανα γιατί θεωρώ ότι ακριβώς αυτό αναμένουν οι πολίτες μας, δηλαδή εργασία και ασφάλεια. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση Θέλουμε μία ανταγωνιστική οικονομία έτσι ώστε οι επενδυτές να επενδύσουν γιατί θεωρώ ότι η εργασία δημιουργείται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και εμείς ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε οι ΜΜΕ να τύχουν χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τις υποδομές την καινοτομία ΜΜΕ, αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, ιδιαίτερα των νέων. Και γι' αυτό το πρόγραμμα που επιθυμούμε μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και του ΣΕΦ και του ΚΟΣΜΕ για τις ΜΜΕ είναι να ενισχύσουμε την όλη διαδικασία ε, στήριξης στο Εράσμους. Δεν, δείχνει, δεν αφορά μόνο τους νέους που ταξιδεύουν. Όταν ε, κάποιος νέος προσλαμβάνεται κάπου, έχει μεγάλη σημασία να έχει διεθνή εμπειρία και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εράσμους, το οποίο υποστηρίζει τους νέους να αρχίσουν καλύτερα τη ζωή τους. Και η πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω, χρειάζονται περισσότερα χρήματα, γιατί η ανεργία των νέων είναι ένα ζήτημα και θα πρέπει να βελτιώσουμε την προτεραιότητα για την πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων. Ως προς την ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, στην κεφαλίδα 3 και 4 είδαμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση τα τελευταία τρία χρόνια. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε κάτι με τα περιορισμένα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους οργανισμούς της Ένωσης που είναι υπεύθυνε ε, για τα εσωτερικά ζητήματα ε, και την εσωτερική τάξη. Αυτό αφορά την ΕΑΖΟ, τη Frontex και άλλους οργανισμούς ε, να έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών ιδιαίτερα για τους ύποπτους τρομοκρατίας, λαθρεμπορίου και διακίνησης ανθρώπων και να ενισχύσουμε και τα εξωτερικά μας σύνορα. Υποστηρίζω και την προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να δαπανούμε 28 φορές τα ίδια χρήματα για την άμυνα. Καλύτερα να δαπανηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να μοιραστούμε τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ως προς την άμυνα και η ασφάλεια στην Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η άμεση γειτονία μας, δηλαδή και η ανατολική ε, πολιτική, πολιτική στα ανατολικά σύνορα, γιατί προς Ανατολάς βλέπουμε μια πιο δραστήρια ομοσπονδία της Ρωσίας και αυτό αφορά και τη Βόρειο Αφρική και την μεταναστευτική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ρίζες της μετανάστευσης και να προβούμε σε, σωστή, σε σωστές δαπάνες. Είναι πολύ πιο εύκολο να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στον τόπο τους. Αυτό είναι πολιτικά πιο εύκολο και όχι τόσο δαπανηρό. Μπορούμε λοιπόν να τους στηρίξουμε περισσότερο εκεί παρά να τους έχουμε εδώ και είναι και πιο ασφαλές. Αυτό αφορά τις δύο βασικές προτεραιότητες. Η δική μου έκθεση για τις κατευθυντηρίες γραμμές ασχολείται με τις κλιματικές αλλαγές επίσης και θα πρέπει να καταβάλουμε και προσπάθεια για να δώσουμε ένα 20% των πόρων στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, στην έκθεσή μου για τις κατευθυντήριες γραμμές ορίζουμε και το πρόγραμμα LIFE, το οποίο θα πρέπει να τύχει στο στις χρηματοδότησης του χρόνου. Και αυτό αφορά και τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμων. Σε σχέση με τους αντίστοιχους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό μας όπως αφορά την ε, ΕΦΣΑ ή βασίζονται σε αυτό χρηματοδότηση όπως ισχύει με τον οργανισμό χημικών ουσιών ή φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμείς θα πρέπει στο μελλοντικό μας προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό 18, να έχουμε προσδώσει τα κατάλληλα κονδύλια, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο στόχο τους. Έγινε λόγος για μείωση του προσωπικού όλων των οργανισμών κατά 5% στο παρελθόν και σε αυτή την περίπτωση μάλλον οι οργανισμοί που άπτονται της δικής σας Επιτροπής και έργου εμπίπτουν σε αυτό το 5%. Στο ε, παρελθόν όλοι έπρεπε να μειώσουν το προσωπικό κατά 5%. Αλλά στη συνέχεια έπρεπε να αυξήσουμε το προσωπικό της Frontex. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε μία κατά περίπτωση προσέγγιση και εκεί που χρειάζονται αυξήσεις θα πρέπει να γίνουν και τούμπαλιν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων βρίσκεται στο Λονδίνο. Θα πρέπει να φύγει από το Λονδίνο όταν αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία. Εμείς θεωρούμε ότι το κόστος αυτό δεν θα πρέπει να το υποστούμε εμείς, ο προϋπολογισμός μας δηλαδή, γιατί δεν ήταν δική μας επιλογή η αποχώρηση της, Ευρωπαϊκής, ε, του, της Μεγάλης Βρετανίας, με συγχωρείτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018 η Μεγάλη Βρετανία θα είναι ακόμα μέλος και γι' αυτό ο οργανισμός θα λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά μετά θα πρέπει να μετεγκατασταθεί και αυτό θα πρέπει να το προετοιμάσουμε. Μιλήσατε για τα πιλωτικά σχέδια και την προπαρασκευαστική δράση της ΕΜΒΗ. Ξέρετε ότι γενικώ η συγητής έχει εύκολο έργο εάν δεν προετοιμάστε πολλά πιλωτικά σχέδια, αλλά εγώ σας ενθάρρυνα να υποβάλετε πιλωτικά σχέδια. Αυτό μου δυσχεραίνει τη ζωή αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερα γιατί θα έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα δεδομένων. Όπως είπε και η πρόεδρος, η ΕΜΒΗ υπέβαλε τα πιλωτικά σχέδια στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και τώρα τα προστέλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια προκαταρκτική αξιολόγηση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε το βαθμό α και να χρηματοδοτήσουμε και τα σχέδια που έχουν λάβει ε, β, αλλά όχι γ, όπως ίσχυσε και πέρσι. Γιατί είχαν χρηματοδοτηθεί τα σχέδια που είχαν λάβει α ή β ως βαθμολογία αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πάντα πολύ ενδιαφέροντα πιλωτικά σχέδια. Αυτό είναι τα σχόλιά μου. Θα ήθελα η παρουσία μου εδώ να σταθεί απαρχή της συνεργασίας μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού κατά τα τέλη Μαΐου και αναμένω και τα δικά σας σχόλια θα αποσταλεί η γνωμοδότηση ως επιστολή, αλλά και το φθινόπωρο θα ήθελα να παραμείνουμε σε επαφή και να μου πείτε με βάση τις πληροφορίες σας ποια είναι τα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα για να τύχουν επαρκούς χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουρασάν. Είσαστε ο εισηγητή της Επιτροπής ε, για τον Προπλογισμό, γι' αυτό και τοποθετηθήκατε στην αρχή. Αυτά που ακούσαμε από εσά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γιατί θίξατε ορισμένα από τα θέματα που μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω και πάλι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για δράσει που έχουν σχέση με το κλίμα, με την βιοπικιλότητα ή με προγράμματα όπω ε, είναι το πρόγραμμα LIFE και ο Μηχανισμός Προστασίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκ μέρους της Επιτροπής μας, θέλω να επισημάνω ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα όσον αφορά τους ε, περιορισμούς του προπολογισμού σχετικά με τις ε, με τους αποκεντρωμένους ε, οργανισμούς. Αν πάρουμε πάνω χάνει τον οργανισμό ή το γραφείο, θέλετε, για το περιβάλλον, ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε προσθέσει πάρα πολλούς ε, κανονισμούς ε, που πρέπει το γραφείο αυτό να τους υιοθετήσει, αλλά παρόλα αυτά ζητάμε μείωση κατά 5%. Άρα δηλαδή κατ' ουσίαν ζητάμε περισσότερη δουλειά, καλύτερη ποιότητα, αλλά με δημοσιονομικούς περιορισμούς. Κάτω από αυτό το πρίσμα ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το γραφείο, να ανταπεξέλθει στα προβλήματα του προπολισμού. Έχουμε και έναν άλλο, ένα άλλο οργανισμό για την ασφάλεια των τροφίμων, πολύ σημαντικός αυτός για τους πολίτες και ίσως θα πρέπει να δούμε λιγάκι τις ε, δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και τους κανονισμούς που ισχύουν έτσι ώστε να ε, μπορούν να λειτουργήσουν πάνελ εμπειρογνωμόνων, να ανατίθενται μελέτες ε, για να ερευνώνται πολλές ε, ουσίες ε, που δημιουργούν ανησυχία στους πολίτες. Κατόπιν υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και όπως είπατε ανησυχούμε διότι θέλουμε να είναι πλήρως λειτουργικός αυτός ο οργανισμός ε, θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην ποιότητα και τη λειτουργία αυτού του οργανισμού που θα μετατεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Παρόλα αυτά, αν λέτε ότι τα κονδύλια για να μετακινηθεί ο οργανισμός αυτός δεν θα πρέπει να προέλθουν από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό γιατί δεν είναι δική μας η υπηρετιότητα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να έχουμε και μια εναλλακτική λύση. Διότι ας μην ξεκινήσουμε με αυτή τη διαφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για το ποιος ε, θα τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά. Και βεβαίως ε, ανησυχούμε και για τα συμβόλαια αυτής της, αυτού του οργανισμού Νομίζω όλα αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά σε σχέση με τη μετακίνηση του οργανισμού. Αυτά καταρχήν είχα να σας πω και βεβαίως ε, θα ήθελα να καλέσω άλλους ε, συναδέλφους, τους και οδησηγητές και άλλα μέλη να λάβουν το λόγο και να εκφράσουν αυτά που τους ε, ενδιαφέρουν. Κύριος Πόρτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, συμφωνώ μαζί σας ε, με αυτά που είπατε και θα ήθελα να υπογραμμίσουμε ένα πράγμα που το... δεν τον έφερε ο κύριος Μουρασάν. Βεβαίως συμφωνώ ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη ενδιαφέρονται για την ασφάλεια, για τις απασχόλησης και για την ασφάλεια όμως, για την ασφάλεια ε, ασφάλεια όχι με την στρατιωτική έννοια, ασφάλεια που είναι σημαντική για τους καθημερινούς, ε, τους απλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, θέλω να το αναφέρω αυτό, ε, πρέπει να έχουμε κατά νου τρία πράγματα. Καταρχήν όταν μιλάμε για το περιβάλλον πρέπει να μιλάμε και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό εκφράζεται μέσα από τον προπολογισμό. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη στρατηγική ε, προκαταρκτικά μέτρα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε όταν θα εμφανιστούν τα προβλήματα που θα εμφανιστούν έτσι και αλλιώς. Ε, διότι νομίζω ήταν το 2011 που εγώ ήμουν σκιώδης ηγητή ε, για τη Λευκή Βίβλο σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλά έκτοτε, ως εκ τούτου θα πρέπει κάπως να επιταχύνουμε, γιατί αν αποτύχουμε αυτό δεν θα είναι καλό για τους πολίτες μας. Το δεύτερο, μιλάμε και για μια άλλη πτυχή της ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, το είπε αυτό και η πρόεδρος, ε, ενδιαφέρονται και για τη χρηματοδότηση των οργανισμών. Δηλαδή στους οργανισμούς φορτώνουμε όλο και περισσότερη δουλειά και τους ε, δίνουμε όλο και λιγότερα χρήματα. Αυτό όμως δεν είναι καλό. Ε, βεβαίως αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι η άποψη της πολιτικής μου ομάδας, αλλά σε τελική ανάλυση δεν ξέρω κατά πόσον ε, ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων μπορεί πράγματι να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Κατόπιν ε, πρέπει να μιλήσουμε για την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας, για τα φυτοφάρμακα, για τον έλεγχο, τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων. Δεν ξέρω κατά πόσον οι έλεγχοι γίνονται ικανοποιητικά. Όλα αυτά πρέπει κάπως να ληφθούν υπόψη. Και όσον αφορά στην υγεία, Σύντομα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε άλλο ένα πρόβλημα που είναι η βακτηριακή αντοχή. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, τα προκατακτικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της βακτηριακής αντοχής απευθύνομαι σε εσά για να μας πείτε πώς ακριβώς ε, θα περιλαμβάνονται αυτές οι προότητες, ε, προτεραιότητες στον προπολογισμό και αν ε, περιλαμβάνονται, γιατί κατά δική μας άποψη δεν περιλαμβάνονται ικανοποιητικά αυτές οι προτεραιότητε στον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σέχαρτ, είναι ένας άλλος και ηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σίγκφριντ, που ήρθε. Χαίρομαι που παίζεις και αυτό το ρόλο και έρχεσαι με αυτή την ιδιότητα εδώ. Πέρα από αυτά που ακούσαμε από την Πρόεδρο και από τον Μπάβελ για τους οργανισμούς, με τα οποία ε, συμφωνώ, ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τις δαπάνες για το κλίμα. Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι 20%. Η Κομισιόν κοιτάει τα νούμερα, κοιτάει πώς γίνονται αυτές οι δαπάνες για το κλίμα σε αυτή τη φάση και έφτασε στο νούμερο του 17%. Λίγο μου φαίνεται. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των δαπανών για το κλίμα τα τελευταία χρόνια ε, πρέπει να είναι πολύ ψηλό, ούτω ώστε να φτάσουμε σε μέσο όρο στην εφταετία στα 20%. Στο 20%. Ε, ορισμένοι με βάση υπολογισμού λένε ότι θα πρέπει να ε, αυξηθούν οι δαπάνε για το κλίμα στο 22% για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέσο όρο. Ε, αυτό το αναφέρετε στην έκθεσή σας, αλλά πολύ γενικόλογα αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν δύο λόγια, πιο συγκεκριμένα, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα έχει δαπανίσει αυτό το 20% ε, για το κλίμα ε, μέχρι το τέλος της ευθετίας. Και επίσης το συμπλήρωμα πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αν διαβάσατε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, μας λέει ότι υπάρχει ένα επιπλέον. Αλλά θα πρέπει εμείς στο Κοινοβούλιο να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να κάνουν περισσότερα πράγματα, για να είναι αξιόπιστοι απέναντι στην ε, συνθήκη του Παρισιού, να δαπανίσουν αυτά που πρέπει. Είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου αυτός νομίζω. Ε, εσύ, Ζίκφριτ, πώς το βλέπεις, πώς ε, θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει η ίδια για τον εαυτό της. Καλό θα ήταν να τους υλοποιήσει εφόσον τους έθεσε η ίδια. Ευχαριστώ κύριε Έκχαρτ. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Σάφετ Πύρικ. Συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε για αυτή τη στρατηγική. Λάβαμε και τα αποτελέσματα ε, την περασμένη εβδομάδα για την Κομισιόν, για το fitness check, για τον έλεγχο καταλληλότητας και για την οδηγία για, το, για τα ενδιατήματα, οικοσυστήματα. Εμείς στην Ολλανδία Ξέρουμε ότι θα υποδεχθούμε την Κομισιόν ε, και θα κοιτάξουμε ένα συγκεκριμένο project, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ε, ότι θα επιλύσουμε τα προβληματικά σημεία. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε τις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά να τις προσαρμόσουμε. Και γιατί το θέτω αυτό, γιατί στη Γαλλία και στον Ομένο Βασίλειο πολλοί από τους ψηφοφόρους λένε ότι αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την παρουσία μας και να δούμε ποια είναι τα προβληματικά σημεία και να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Ε, ανησυχώ επίσης για τις οικονομικές δραστηριότητες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αλλά και την ειδική ρήτρα και την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Πολύ ωραία. Ακούσατε όλους τους ευρωβουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Ε, ο λόγος σε εσάς κύριε Μόρεσαν. Καταρχά, για τι δικέ σα παρατηρήσει για του οργανισμού. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντο να αποτελέσει ένα κλασικό παράδειγμα, είναι μάλλον ένα κλασικό παράδειγμα, όπου ο στόχος του 5% που εφαρμόστηκε σε όλους τους οργανισμούς ήταν εντελώς ακατάλληλος, γιατί είχε όλο και περισσότερα καθήκοντα, λιγότερα λεφτά. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά για το μέλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το έργο της κάθε υπηρεσίας, του κάθε οργανισμού. Και το ο γενικός κανόνας είναι ότι όσοι λαμβάνουν περισσότερες αρμοδιότητες θα πρέπει να έχουν και περισσότερο, μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων και μεγαλύτερο προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ε, δεν θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε τη μετακατάστασή μας. Ε, είναι ένας οργανισμός της Ένωσης. Ε, η λειτουργία της θα πρέπει να ε, εξασφαλιστεί απρόσκοπτα, δεν θα πρέπει να πέσει θύμα του Brexit. Εξυπηρετεί τώρα 28 κρατη και μετά θα εξυπηρετεί 27, ανεξάρτητα από το πώς θα λάβει η χώρα το Brexit. Γι' αυτό μαζί σας είμαι και εγώ. Συμφωνώ δηλαδή ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός φαρμάκων θα λειτουργεί και θα λειτουργήσει, ανεξάρτητα από το που θα πάει και πότε θα, θα μετεγκατασταθεί από το Λονδίνο. Επίσης, με ρωτήσατε για τις δαπάνες, για τους α, κλιματικούς στόχους. Το πώς θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, δηλαδή, κτλ. Έχεις δίκιο έχουμε καθυστερήσει. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η αναθεώρηση του εφταετούς προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το 2013 συμφωνήσαμε για το δημοσιονομικο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Όταν το συμφωνήσαμε, πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, τρομοκρατία, έλλειψη ασφάλειας, μετανάστευση, δεν τα είχαμε προβλέψει το 2013 χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα λεφτά που βρήκαμε κάπου στον προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε την ε, προσφυγική κρίση. Σωστό ήταν αυτό και χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμω, ε, η εφταετία είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνήσαμε το Συμβούλιο όταν δια... διαπραγματευτήκαμε την αναθεώρηση ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Θα έπρεπε να υιοθετήσουμε την αναθεώρηση την περασμένη εβδομάδα έπρεπε να την υιοθετήσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ε, αλλά δυστυχώ το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε λόγω των εκλογών να καθυστερήσει την υιοθέτηση. Δεν είπα ότι μπλοκάρουν την υιοθέτηση τη αναθεώρηση του πλαισίου, αλλά την αναβάλουν. Δύο ή τρει μήνε θα την αναβάλουν λόγω των εκλογών, λένε. Ε, αυτό θα μα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, αν γίνει τότε, μέχρι τέλο ε, Ιουνίου. Αν όμω δεν υιοθετηθεί η αναθεώρηση αυτή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λεφτά ε, σε τομεί που δεν είχαμε προβλέψει ότι θα είναι προβληματική το 2013. Και είναι οι τομεί όπου έχουμε καθυστερήσει πραγματικά. Ακριβώ λοιπόν η απάντηση βρίσκεται εκεί. Η αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι μια ανοιχτή πόρτα για μας. Δηλαδή, μας δίνει ευελιξία, θα μας δώσει αυξημένο προπολογισμό στους τομείς που τον χρειαζόμαστε και έχεις πολύ δίκιο ότι θα χρειαστεί μια ενιαία θέση από το Κοινοβούλιο, μια κοινή προσπάθεια από πλευρά μα για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Όταν λέω να πιέσουμε τα κράτη-μέλη όμω, ξέρω πολύ καλά ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ξοδεύουμε τα ποσά που προβλέπει ο προπολογισμό στην ΕΤΑ. Για κάθε ευρώ που δαπανάτε θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Απλά. Ε, αυτά. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική υπευθυνότητα. Αυτό είναι σημαντικό, το θέλουν και οι πολίτε. Αλλά αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε νέε προτεραιότητες χωρί νέο χρήμα, χωρί φρέσκο χρήμα, πώ θα γίνει, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ θα πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι αν μας ζητηθεί να κάνουμε πολύ περισσότερα με τον προπολογισμό που αποφασίστηκε το 2013 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επομένω σε κάποιου τομεί θα πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση. Αυτά έχω να σας πω εγώ για τη βιοπικιλότητα. Υπάρχει στις κατευθυντήριες γραμμές μου ότι δυστυχώς ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ε, δεν θα υλοποιηθεί χωρίς ουσιαστικές προσπάθειες. Τονίζουμε επίσης τη σημασία απλούστευσης της προστασίας της βιοπικιλότητας και της ένταξης στον προϋπολογισμό του θέματος αυτού. Ε, εστιάζουμε κυρίως ε, στο δίκτυο Natura 2000 και στο LIFE όταν του χρόνου κάνουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Το Μάρτιο, ή μάλλον δεν την κάναμε το Μάρτιο, ο Έτιγκερ είπε ότι δεσμεύεται να ενσωματώσει όλα, όλα όσα έχουμε βάλει στις κατευθυντήριες γραμμές μας. Θα πρέπει όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε σε αυτό που θα μας παρουσιάσει η Κομισιόν τέλος Μαΐου και με αυτή την έκθεση στα χέρια μας θα πρέπει από κοινού να πιέσουμε ακόμα περισσότερο του την Κομισιόν. Αυτό εν μέρει απαντάει και την ε, ερώτηση που έθεσε ο κύριος Πότς. Δηλαδή, όταν η Κομισιόν ετοιμάσει το προσχέδιο προπολογισμού το, στα τέλη Μαΐου, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε μονοσήμαντα τις προτεραιότητες, τις αρχές, τις πολιτικές προτεραιότητες και να δούμε τα νούμερα αυτή στιγμή Μα προτείνει η Κομισιόν τέλο Μαΐου με το προσχέδιο του προπολογισμού τα δικά τη νούμερα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε επαφή και γι' αυτό Πρόεδρε, θα περιμένω την επιστολή που θα στείλετε στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα τη λάβω υπόψη μου. Και σας ευχαριστώ βεβαίως για την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη δουλειά σας και για τη δέσμευσή σας να λάβετε πολύ προσεκτικά υπόψη τα πιλωτικά προγράμματά μας. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πολλές καλές ιδέες αυτά και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που έχετε εκφράσει ήδη από τώρα. Ευχαριστώ και καλό απόγευμα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που έχει σχέση με την μέρημνα υγεία σε διασυνοριακά και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή ΡΙΣ. Ξεκινάμε λοιπόν ε, κύριε Διευθυντά, με εσά, με τα σχόλιά σας και μετά θα επανέλθω στους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για αυτή την οδηγία, τη διασυνοριακή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή η οδηγία ήταν κάτι το πολύ επιτυχημένο σχετικά με την πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε το 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και άρχισε να εφαρμόζεται το 2013. Ο στόχος, η πολιτική αυτή είχε στόχο καταρχήν τη διασυνορική ε, μέρημνα υγείας. Έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο για να προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες ε, στα εθνικά <laughs> συστήματα υγείας και επίσης η οδηγία αυτή επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, υπάρχει συνεργασία σε μία σειρά θεμάτων τα θέματα τα οποία, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε δείχνουν ότι υπάρχει μια σειρά ασθενών οι οποίοι μετακινούνται και θα μετακινούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ας δούμε λιγάκι την εφαρμογή της οδηγίας. Από τότε που εγκρίθηκε η οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει το κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η οδηγία από τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εργαζόμαστε στα περίφημα ε, check ε, συμμόρφωση, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε πώς ακριβώς αυτή η οδηγία μεταφράζεται και ενσωματώνεται στα εθνικά συστήματα. Μιλάμε για την οδηγία, για ένα νομικό εργαλείο και τα κράτη-μέλη προφανώς και έχουν κάποια ευελιξία στην μεταφορά αυτή τη οδηγία στην εθνική του νομοθεσία. Κυρίω γιατί μιλάμε για διαφορετικά συστήματα υγεία για διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ε, καλύπτεται χρηματοδοτικά υγεία, διαφορετικέ διατάξει. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία ε, στα δικά τους ε, τα νομοθετικά συστήματα, αλλά η Κομισιόν κατ' ουσίαν παρακολουθεί την κατάσταση ε, και κυρίως επεμβαίνει οποτεδήποτε δεν εφαρμόζεται η οδηγία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπανά χρόνο και προσπάθειες για να εντοπίζει παραβιάσεις του κοινωτικού δικαίου που επηρεάζουν την υγεία των ασθενών. Υπάρχουν ειδικέ περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά αυτή την οδηγία και θα αναφέρω δεικτικά κάποιους τομείς που εξετάζουμε. Πρώτον, όσον αφορά τις επιστροφές για θέματα δαπανών υγείας, κατόπιν ε, το θέμα της τιμολόγησης για ασθενείς από άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε μακροσκελείς καταλόγους ε, που απαιτούν ε, την εξοδότηση και τελικά υπάρχουν διαφορετικές ε, νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην επιστροφή δαπανών. Υπάρχει και ένα θέμα που έχει σχέση με το ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια ζημιά εις βάρος των ασθενών. Οι Κομισιόν ε, έχουν γίνει λοιπόν πάρα πολλές ε, συζητήσεις και προσπαθούμε να ζητήσουμε μια καλή λύση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το εξής. Λόγω αυτής της ύπαρξης αυτής της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, προφανώς και επικαιροποιούμε αυτή την έκθεση και πρόκειται να καταθέσουμε και μία έκθεση η οποία έκθεση θα κατατεθεί ε, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τον Οκτώβρη του 2018. Ως εκ τούτου έχει ήδη ξεκινήσει η όλη διαδικασία και θέλουμε να δείξουμε, να μπορέσουμε τότε να δείξουμε πώς ε, εφαρμόζεται αυτή η οδηγία στα τρία χρόνια που ισχύει, να έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα. Επίσης, έχουμε χαρτογραφήσει διαδικασίες ε, διασυνοριακές σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες, στα κράτη-μέλη. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα διασυνοριακά προγράμματα. Επίσης, γίνονται μελέτες για να εντοπίσουμε checklists ε, για τις ε, τοπικές κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, το πώς μπορεί στο μέλλον να ε, οργανωθεί η συνεργασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να οργανώσουμε και μία μελέτη για να διαπιστώσουμε την ε, διαθεσιμότητα πληροφοριών στους ε, ασθενείς που προσπαθούν να νοσηλευτούν και με διασυνοριακές υπηρεσίες. Η έκθεση είναι μια πολύ καλή έκθεση γιατί καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις, τα μέτρα τα οποία προτείνει η οδηγία. Ελπίζουμε λοιπόν Όλη αυτή η διαδικασία με πάρα πολλέ μελέτες, αξιολόγηση, εκθέσει ε, που έρχονται από τα κράτη-μέλη και από ανεξάρτητους συμβουλευτικού οργανισμούς. Ελπίζουμε ότι με όλα αυτά θα έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το πώ ακριβώς εφαρμόζεται η οδηγία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε την τελευταία φορά που συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο ήταν η συνδυτοποίηση. Όπως ε, λοιπόν ε, δείχνει το ευρωβαρόμετρο το ότι υπάρχουν αυτά τα νέα δικαιώματα για τους ασθενείς, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα συνειδητό, δεν έχει διαδοθεί και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να διαδώσουμε περισσότερες πληροφορίες και στους ασθενείς και στις οικογένειές τους για να γνωρίζουν τις υπηρεσίες υγείας διασυνοριακά. Ένα κρίσιμο εργαλείο που έχουμε στην οδηγία και στη συνεργασία με την ακρατημέλη είναι τα εθνικά σημεία επαφής τα οποία σημεία αυτά παίζουν πολύ σημαντικό καθοριστικό ρόλο γιατί προσφέρουν ε, υπηρεσίες, πληροφορίες στους ασθενείς, ε, στις οικογένειές τους, εφόσον βέβαια τους ζητηθεί και καλούνται αυτά τα σημεία ενημέρωσης να προσφέρουν ε, τις πληροφορίες στους πολίτες των κρατών μελών, αλλά να επικοινωνούν τα σημεία αυτά και μεταξύ τους. Όσον αφορά στη συνειδητοποίηση και ενημέρωση για την οδηγία, τον Οκτώβριο που μας πέρασε οργανώσαμε μία ε, συνδιάσκεψη για να ενημερώσουμε και για να είναι γνωστό ότι μπορούν διάφοροι φορείς να συζητήσουν για το πώς μπορούμε να ε, επικοινωνούμε με τους ε, πολίτες. Επίσης για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σχέση με τους επαγγελματίες της ε, υγείας, να μπορούν και οι επαγγελματίες να προσφέρουν ε, υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς από άλλες χώρες. Τώρα, να πω και λίγα λόγια για το πώς λειτουργούν όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη. Όσον αφορά στα εθνικά σημεία επαφής, στην ε, έκθεση ε, με την βοήθεια των κρατομελών μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία και λάβαμε πληροφορίες ε, για περίπου 60.000 πληροφορίες που μπορούν να ανακληθούν από τα σημεία ενημέρωσης και επαφής. Μπορούν να ανακληθούν και μέσω Skype, αν είναι αυτό απαραίτητο. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η χώρα η οποία προσφέρει πολλές πληροφορίες στους ασθενείς είναι η Πολωνία. Και επίσης αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι τα σημεία επαφής ε, και επικοινωνία στη χώρα αυτή χρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αυτά τα εθνικά σημεία επαφής, έρχει, οργανώνει συναντήσεις, ε, στηρίζει μελέτες που αφορούν ε, στη δουλειά τους και μάλιστα αυτή την Παρασκευή θα ξανασυναντηθούμε για να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εθνικά σημεία επαφής και να συζητήσουμε και για την εμπειρία τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει κατανοητό το πώς αλλάζει η επικοινωνία και το ότι πρέπει να γίνουν μελέτες σε βάθος για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι τρέχουσες ανάγκες ε, των ασθενών, των οικογενειών τους, αλλά και των επαγγελματιών της υγείας. Νομίζω λοιπόν ένα πολύ πετυχημένο κομμάτι αυτής της οδηγίας είναι εκεί που γίνεται λόγος για τη συνεργασία Το Κοινοβούλιο το γνωρίζει αυτό. Πρόσφατα ε, εισαγάγαμε ε, δίκτυα επαφής και βλέπετε και μία εικόνα από τη συνάντηση στο Βίλνιους αρχές Μαρτίου όπου πιστοποιήθηκαν 24 δίκτυα από τον Επίτροπο Αντρουκάητης. Αυτό πραγματικά ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Ευρώπη. Ε, οι άνθρωποι συναντήθηκαν κορυφαίοι γιατροί της Ευρώπης από 313 νοσοκομεία, από 25 κράτη-μέλη, από 950 κλινικές. Όλοι αυτοί πρότιμοι να συνεργαστούν και αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η ψηφιακή υγεία, ηλεκτρονική και ψηφιακή υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ηλεκτρονική αυτή μορφή παροχής υπηρεσιών υγείας, γιατί ο στόχος είναι να προσφέρονται λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν σε καλύτερη υγεία και να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει συνεργασία, τακτική συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις ε, κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Γιατί αναπτύσσουμε, φτιάχνουμε ένα πολύ σημαντικό πόρταλ, μια πύλη ε, στο πλαίσιο του Connecting Europe. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η αξιολόγηση της τεχνολογίας που υπάρχει για την υγεία ε, το Κοινοβούλιο προτίθεται να προτείνει πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη συνεργασία μέχρι τα τέλη αυτού του έτους. Αυτή λοιπόν η μορφή συνεργασίας είναι εφικτή λόγω της ε, διάθεσης ε, της, των κρατών μελών αλλά και λόγω της συνεργασίας με το πρόγραμμα UNETA είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, και ενεργός ο ρόλος που παίζουν διάφοροι εμπλεκόμενοι και φορείς ε, στον τομέα αυτό. Και τέλος, ε, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει και μία ανακοίνωση για συνεργασίες που θα διαμορφώνονται. Εμείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία και να παρουσιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Τελειώνοντας, ήθελα να πω κάτι που ανέφερε ο επίτροπο μου, ο οποίος είπε ότι αυτή η οδηγία είναι ρηξικέλευτη, είναι μια χρυσή ευκαιρία για να δείξουμε τα ευρωπαϊκά ωφέλη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να τύχει εκμετάλλευση, πλήρω εκμετάλλευση, το δυναμικό που υφίσταται. Ε, σας ευχαριστούμε και πρέπει να δώσουμε καταρχάς ε, το λόγο ε, στην κυρία Γκολστέτ που είναι η συγγήτρια για την οδηγία αυτή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την Κομισιόν που ε, μας ξαναμιλάει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Να υπενθυμίσω για τους συναδέλφους που ήταν τότε στο παρελθόν ε, όπου χρειάστηκε να δουλέψουν πάνω σε αυτήν την οδηγία ότι είναι περήφανο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καταλήξαμε σε ένα τέτοιο κείμενο για τη διασυνοριακή περίθαλψη και έχουμε εδώ την ε, αναμφισβήτητη απόδειξη τα, για τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε όταν συνεργαζόμαστε παρά όταν δουλεύουμε μεμονωμένα. Μιλήσατε για το πώς εξελίχθηκε η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Να σας υπενθυμίσω ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τότε στο παρελθόν, την απροθυμία που συναντήσαμε από πλευράς κατών μελών για να δεχτούν την ύπαρξη αυτής της οδηγίας. με βάση αυτά που μας είπατε, βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά που, που πρέπει να γίνουν. Δεν θα πρέπει να παρετηθούμε, γιατί ξέρουμε τις τροχοπέδες που βάζουν τα κράτη-μέλη, που έχουν την τάση να βάζουν για τέτοια θέματα. Λοιπόν, πρέπει να υπαγρυπνούμε, μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Μου άρεσε που μας εξηγήσατε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ευαισθησία των πολιτών και να ενημερωθούν για την ύπαρξη αυτής τη οδηγίας. Ε, σημείωσα την πρόοδο που έχει σημειωθεί για το e-health, για την ηλεκτρονική υγεία. Ε, εγώ τότε, ήθελα, στο παρελθόν, ήθελα να σπρώξω για να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Και δυστυχώς χρειάστηκε να κάνω πίσω και να δεχτώ την απλή αναφορά της δυνατότητας αυτής, που ήταν μια μεγάλη καινοτομία, απλώς ε, σε ένα κείμενο. Είχαμε απλώ μια αναφορά για το e-health σε ένα κείμενο. Και τώρα βλέπω ότι επιτέλου όλα αρχίζουν να έτσι, λειτουργούν. Αρχίζουμε να βλέπουμε τη διαλειτουργικότητα που ήταν ε, πραγματικά εκ των ονουκάνευ, ούτω ώστε να προχωρήσουμε για αυτή την ψηφιακή υγεία, ε, δεδομένης και της ε, πρόοδου της τεχνολογίας της υγείας. Ευτυχώς, προχωράμε, ευτυχώς. Αλλά παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο και ευχαριστώ την Κομισιόν για όλα θα κάνει. Υπάρχει ένα βασικό μέτρο που είναι η εφαρμογή των ε, Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς για τις σπάνιες και περίπλοκες ασθένειες. Ε, έχει γίνει πολλή δουλειά και χαίρομαι που δημιούργησα 24 πρώτα, ένα πρώτο κύμα 24 δικτύων για αυτές τις αρρώστιες. Ε, στη δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχουν διάφορα νοσοκομιακά κέντρα που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και μου μίλησαν. Ε, είδα ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από πλευράς πολλών νοσοκομείων. Είναι μια καλή προσπάθεια, είναι πρόοδος, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν πραγματικά αυτά τα ευρωπαϊκά δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ξεκινήσει την πορεία, αλλά σε επαγρυπνούμε, ούτως ώστε να συνεχιστεί η πρόοδος. Επίσης, όταν δημιουργήσουμε αυτά τα δίκτυα αναφοράς, θα βελτιωθούν και η, διάγνωση, και, το, και η διάγνωση, αλλά θα μπορέσουμε να αναλάβουμε και να δώσουμε θεραπεία στους ασθενείς με σπάνιες αρρώστιες, από όπου και αν προέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να βάλουμε από κοινού τα μέσα που έχουμε. Και αυτό θα μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος. Θα πρέπει να ενημερώσουμε για την ύπαρξη αυτών των δικτύων. Θα πρέπει οι πολίτες και οι ασθενείς να μάθουν αυτά τα δίκτυα. Θα πρέπει να διευκολύνουν τους ασθενείς που θέλουν να έχουν πρόσβαση και όσους θέλουν κυρίως να πάνε στο εξωτερικό. Μας είπατε ότι πάνω από 60.000 αιτήσει ενημερωτικές ε, κατατίθεται στα εθνικά ε, σημεία επαφής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους πολίτες μας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όμως τα οποία είναι έτσι εκρεμή. Η κατάσταση από κράτο μέλο σε κράτο μέλο διαφέρει πολύ σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτών των εθνικών σημείων επαφής. Η αποτελεσματικότητα και οι αρμοδιότητε που έχουν είναι τελείως διαφορετικέ από κράτο σε κράτο. Ε, θα πρέπει όμως οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση, να, είναι, ε, να αντιμετωπίζονται ισότιμα απέναντι στα επίγοντα προβλήματά τους. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι η Κομισιόν και το Κοινοβουλίο θα πρέπει να συνεργαστούν οπωσδήποτε, ούτως ώστε να υποχρεώσουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς το συμφέρον των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Συνάδελφοι, εάν θέλετε να μιλήσετε για το θέμα αυτό, θα σηκώσετε το, το χέρι σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσυπογράφω αυτά που μόλις προανέφερε η κυρία Γκροστέτ. Αν μιλάμε για μεγαλύτερη διαδικασία συνειδητοποίησης, υφίσταται αυτή, αλλά υπάρχουν και στενοποί σε σχέση με την διαδικασία χρηματοδότησης, γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικά συστήματα υγείας και ο ασθενής δεν ξέρει πώς πρέπει να προχωρήσει. Όταν πρόκειται για το καθεστώς προαδειοδότησης, σε περίπτωση δηλαδή ατυχήματος στο εξωτερικό, πρέπει να πάει κανείς στον γιατρό που τον παρακολουθεί, μα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να το επεξηγήσουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος ε, των νοσηλείων, της περίθαλψης και, όλα τα και ούτω καθεξής. Στην Ολλανδία, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της χώρας, είναι δυνατόν να λαμβάνουμε πιο εύκολα αυτή την προαδειοδότηση, ιδιαίτερα στο Γκρένιγκεν, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή για αυτή την έκθεση, καθώς και την κυρία Γκροστέτ. Πράγματι, εμείς ως θεσμικό όργανο αλλά και η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ περισσότερα για την πρόσβαση στα εθνικά συστήματα υγείας όταν ε, μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την προστιθέμενη αξία για τους πολίτες. Ως προς την οδηγία, θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε στους ασθενείς ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια των περιορισμένων αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων. Θέλουμε όμως να ε, βελτιώσουμε την ε, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι η επίπτωση της οδηγίας σε σχέση με την υγειονομική περίθαλψη και τις ανισότητες. Υπάρχει εν τη γενέση ένα σχέδιο για να έχουμε δείκτες υγείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις ανισότητες στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιπτώσεις της οδηγίας για να μειωθούν οι ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην ε, περιθάλψη. Η κυρία Ντορνάτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη οδήγησε στον ιατρικό τουρισμό. Στην Ευρώπη μιλάμε για ένα 4% το 2016, δηλαδή 46 δις ευρώ. Η οδηγία αυτή οδήγησε σε έναν ανταγωνισμό και σε μία εξειδίκευση των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να μην δεχτούμε αυτή την κινητικότητα όταν πρόκειται για σπάνιες ασθένειες ή για ειδικέ τεχνολογίες. Όμως αυτή η πρακτική οδηγεί σε μια ιατρική δύο ταχυτήτων. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της περίθαλψης τη στιγμή που οι πρακτικές διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο. Έχετε προβλέψει μέτρα εναρμόνισης ε, της περίθαλψης και ιδιαίτερα σε σχέση με την παρακολούθηση των ασθενών διασυνοριακά. Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μία ομάδα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και επικοινωνίας δημιουργήθηκε για να ε, χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Με αυτές τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου, οι γιατροί ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με τον ασθενή. Θα ενισχύσετε το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Διευθυντή τον κύριο Ρίς, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Όπως γνωρίζετε πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το κόστος περίθαλψης σε ένα άλλο ε, κράτος μέλος. Έχετε μία εκτίμηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Κύριε Ρης, έχετε το λόγο για να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα αναφερθώ στην κυρία Γκροστέτ γιατί μίλησε εκτενώς για τις εξελίξεις στον τομέα. Συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να επιζητούμε και τη συνεργασία των κρατών μελών. Συνεχίζουμε αυτή την εργασία. Έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα με τα κράτη-μέλη σε δύο περιπτώσεις ε, ολοκληρώθηκαν τα σχέδια γιατί τα κράτη-μέλη ήταν συνεργάσιμα και ελπίζω να έχουμε παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλες περιπτώσεις και χώρες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την πίεση αλλά και τη συνεργασία γιατί τα συστήματα είναι τόσο διαφορετικά, δηλαδή ε, οι διατάξεις αυτές της οδηγίας αφορούν ένα ειδικό πλαίσιο εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στα δίκτυα αναφοράς των κρατών μελών. Ήταν ε, χρονοβόρα η διαδικασία σύστασης του συστήματος και προσπαθήσαμε να ε, συνεργαστούμε με τις κλινικές και τους γιατρούς, κάτι το οποίο καταφέρα. Έχουμε 22 δίκτυα αυτή τη στιγμή και ε, δύο δίκτυα είναι ακόμα πιο ε, περίπλοκα. Αφορούν την επιληψία και τις παιδικές μεταμοσχεύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε μέσα στα πλαίσια του δικτύου, αλλά υπάρχουν και άλλοι κλινικοί τομείς. Δεν θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα θέλαμε ε, το 2019 να επεκταθούμε με τα 24 δίκτυα θα αρχίσουμε με τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντας, ενδιαφέροντας από τα κράτη-μέλη για να συνεργαστούν και άλλα κράτη με τα 24 δίκτυα. Αυτό για να απαντήσω στον κύριο Κόβατσεφ. Προσπαθούμε διυπηρωτικά να αναπτύξουμε αυτά τα ε, δίκτυα γιατί μπορεί ένα κράτος να μην προσχωρήσει αυτή τη στιγμή, αλλά αργότερα. Θα υπάρχει η δυνατότητα προσπογραφής. Υπάρχει, υπάρχουν αυστηροί όροι πρόσβασης στο δίκτυο, γιατί θέλουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα τεχνολογικά δίκτυα θα δούμε πώς θα συντονίσουμε τα 24 δίκτυα μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας συνεργασίας. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σύστημα και προωθούμε τη συνεργασία προβάλλουμε ε, λύσεις ε, με βάση του, ε, συνδέοντας, του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, του ΣΕΦ, καθώς και των υποδομών, των νοσοκομιακών υποδομών. Υπάρχει και το πρόγραμμα e-health. Αυτή η συνεργασία κινείται με βάση τις συμφωνίες και την ενιολογική βάση σε κατευθυντήριες γραμμές και μια πραγματικότητα. Ελπίζουμε λοιπόν αν έχουμε πολλά κράτη που θα προσυπογράψουν του χρόνου, θα προβούμε σε ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και ηλεκτρονική συνταγογράφηση Άρα όλοι θα συμμετέχουν στο μεγαλύτερα σύστημα του, την επόμενη χρονιά. Έχουμε ιστορίες επιτυχίας, δεν θέλω όμως να πω ε, πολλά γιατί τώρα μπαίνουμε στην νέα φάση του συστήματος IT. Πρόκειται για, περίπλοκο, για ένα περίπλοκο σύστημα. Θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη τα γλωσσικά ιδιώματα αλλά και τα σημασιολογικά πεδία των γλωσσών, την ε, ιατρική ιδιόγλωσσα και ούτω καθεξής. Ως προς την ε, κατάρτιση των εθνικών φορέων, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, προβούμε σε ανταλλαγή γνώσης ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τη γνώση, με τους ιστότοπους. Να δούμε κατά πόσο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στα δίκτυα ψηφιακής πληροφορίας και πληροφόρησης. Άρα μιλάμε για κατάρτιση και γνωστικό πεδίο. Η κυρία Σάινερ μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αρχική, αρχική μας συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ενεργούνται μελέτες για να δούμε πώς ε, προχωρούμε και με τις συμβατικές σχέσεις για να δείξουμε και στις περιφέρειες πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας υπάρχει στενή συνεργασία όπως και στις όμορες περιοχές της Γερμανίας, το Μπενελούξ. Και φυσικά, όπως είπα, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Βέλγιο συνεργάζονται στενά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη σωστή εργαλειοθήκη για τις περιφέρειες που θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη συνεργασία. Και με βάση αυτή τη μελέτη θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε και να αποβράλουμε μία σύνδεση και με τις γερμανικές περιφέρειες. Ως προς το θέμα της προσβασιμότητας που είπε και ο κύριος Κόβατσεφ, είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε άμεσα ε, να προβάλλουμε αυτή τη συνδεσιμότητα. Υπάρχει μία υποδομή η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους ασθενείς της πόλης και ούτω καθεξής. Δηλαδή η Σόφια μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν νεύρο χειρουργό ε, οποίος, με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή από τη Λιόν, ο οποίος ε, επέστρεψε στη Σόφια και μπόρεσε να χειρουργήσει και να αντιμετωπίσει μια περίπτωση επιληψίας. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτή την οδηγία να ε, οδηγήσουμε στην διακίνηση της γνώσης και όχι των ε, ασθενών. Αλλά φυσικά πολλές φορές πρέπει να μετακινηθούν και οι ασθενείς εκεί που υπάρχουν οι υποδομές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών. Η θεραπεία πρώτων υπάρχει σε ορισμένες χώρες, σε άλλες όχι. Έχει σημασία λοιπόν αυτό. Επίσης και οι γενετικές δοκιμές. Είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρουμε ε, δείγματα για αιματολογικές εξετάσεις παρά να μεταφέρουμε τους ασθενείς. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της ε, διαγνωστικής διαδικασίας γιατί ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα. Δηλαδή μιλάμε για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά σημεία επαφής για να ξέρουν οι ασθενείς που μπορούν να λάβουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Η κυρία Ντορνανό μίλησε για, το, για την κατάρτιση η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβάλλει τις ελάχιστες προδιαγραφές κατάρτισης ιατρικού προσωπικού και αυτό αφορά και τις ΜΕΣ και τα φαρμακεία και ούτω καθεξής. Γιατί η κατάρτιση είναι μέρος της λύσης. Μέσα στα πλαίσια του δικτύου θέλουμε να αυξήσουμε αυτή την ικανότητα κατάρτισης διαμέσου των δικτύων. Έχουμε πολλές, πολύ καλές εξελίξεις από τους ιατρικούς φορείς, ε, έτσι ώστε στους τομείς ε, ουρολογίας, αναισθησιολογίας και άλλων τομέων να μπορέσουμε να αυξήσουμε ε, τις προδιαγραφές και να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο εξετάσεων. Υπάρχουν και μεταπτυχιακές ε, καταρτήσεις. Η Μάλτα τώρα έχει εκκινήσει μια διαδικασία. Θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Μιλήσαμε για γενετικές πληροφορίες κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα και θα φτάσουμε σε νέες εξελίξεις. Πρόσβαση στα δεδομένα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα να μπορούμε να τα μοιραζόμαστε και να έχουν πολύ καλή ποιότητα, γιατί μιλάμε για γενετικές δοκιμές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό έχει σημασία να το δούμε αυτό μέσα στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Ε, δηλαδή να, υπάρχουν, να υπάρχει σωστή συμβουλευτική όταν μιλάμε για γενετικές δοκιμές. Τέλος, η πρόεδρος μίλησε για τα εθνικά πλαίσια τα οποία μπορούν να ενισχυθούν. Συγγνώμη ένα λεπτό. Να δω τις σημειώσεις μου για την εφαρμογή της οδηγίας. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Πιστεύω ότι κατά τα τέλη του 2018 θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της οδηγίας. Υπάρχει βέβαια και το όριο με τον κανονισμό. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς χρησιμοποιούμε και τον κανονισμό για τις κοινωνικές παροχές. Υπάρχει μία σειρά ζητημάτων που σχετίζεται με τα μεμονωμένα εθνικά συστήματα και πώς αντιμετωπίζουν αυτή την οδηγία. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα, αλλά και θέματα. Δηλαδή ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας πούν κατά πόσο υπάρχουν εθνικές δικαστικές υποθέσεις Είχαμε τέτοιες ε, διαδικασίες όπου δεν αποφάνθηκε τελικά το δικαστήριο και νομίζω ότι υπάρχουν και υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά δεν θα ήθελα να προχωρήσω, γιατί βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Αυτή η οδηγία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά από όλους τους συμμετέχοντες. Πολύ σύντομα, γιατί κανονικά δεν προβλέπεται από τη διαδικασία. Μιλήσατε για τις ε, μεμονωμένες χώρες, όπου μερικές φορές η ασφάλεια δεν γίνεται δεχτή. Στο Βέλγιο, ας πούμε, να σας πω, εγώ άρχισα να μου ματώνει μύτη μια μέρα και δεν σταματούσε και η ιατρική υπηρεσία του Κοινοβουλίου με παρέπεμψε σε ένα νοσοκομείο. Εκεί έλαβα θεραπεία. Του έδειξα την μπλε κάρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να πληρώσω μαθή, γιατί ήταν επίγον το θέμα. Και στο Βέλγιο μου είπαν ότι δεν δέχονται αυτή την μπλε κάρτα. Και ήθελα να του πληρώσω ε, τριτά. Δεν ήταν ένα ποσό τεράστιο που δεν μπορούσα να πληρώσω, αλλά φαντάζομαι πως 90 ευρώ ήταν, αλλά νομίζω ότι θα προτιμούσε ένα τουρίστα να χρησιμοποιήσει την ε, μπλε κάρτα και να πληρώσει με αυτή, παρά με ρευστό. Κυρία Γκοστέτε, Ε, υπάρχει η εξή διάκριση. Ορισμένοι πρέπει να δεχτούν ε, θεραπεία κατεπηγόντως και ορισμένοι ε, προγραμματίζουν ας πούμε, την ε, αγωγή τους η οδηγία αυτή ε, για διασυνορική περίθαλψη αφορά τις προγραμματισμένες υπηρεσίες υγείας. Ε, οι κατεπίγουσες ε, υποθέσεις λαμβάνονται υπόψη και τις αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία χωρίς πρώτερη έγκριση. ξέρω ότι δεν πρέπει να μακρηγορήσω, αλλά δεν μπορώ να αφήνω να λένε ότι αυτή η οδηγία ε, προωθεί τον, ιατρικό τουρισμό. Όχι, αντίθετα, για να τον αποφύγουμε γίνεται. Δεν αφορά καθόλου τον ε, ιατρικό τουρισμό. Το σύστημα των πρώτερων ε, εγκρίσεων ακριβώς μας οδηγεί στο να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Θα πείτε στους γονείς, ας πούμε, ενός παιδιού το οποίο πάσχει από ένα σπάνιο καρκίνο ότι χρειάζεται να γίνει μια διάγνωση και ότι δεν μπορεί να υποφεληθεί από, ένα, από τις γνώσεις ενός μεγάλου καθηγητή γιατί είναι σε ένα άλλο κράτος μέλος ή γιατί εκεί που, είναι, που ζουν αυτοί οι γονείς, ε, που μένουν μάλλον αυτοί οι γονείς, δεν υπάρχει αυτός ο, αυτή η γνώση ή εν πάση περιπτώσει αν χρειαστεί να πάνε και να δουν τον καθηγητή οι γονεί, ε, αυτό το ταξίδι θεωρείται ιατρικό τουρισμό, είναι ντροπή αυτό. Είναι λάθο για όλου αυτού που δούλεψαν σκληρά για να υπάρξει αυτή η οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Και πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. Γιατί, Γιατί ο στόχο μα είναι, είναι η ισότητα όλων των πολιτών, όλων των ασθενών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτω ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν όλοι από μια ποιοτική υγεία. Αυτό ήθελα να πω. Thank ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχατε στη συζήτηση. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πού είναι μία αντίρρηση. Προτείνω να τη δούμε μαζί, μαζί με το σημείο 7, 6 και 7 δηλαδή, 5, 6 και 7. Ε, έχουμε το άρθρο 106, Καταρχάς θα πρέπει να εγκρίνουμε το τροποποιημένο ε, βαμβάκι GHB 119 ε, να μπει στην αγορά και το DAS 40 279 γενικά τροποποιημένο αναβόσιτο. Τα 6 και είναι αυτά τα δύο σημεία τα 6 και τα 7. Έχουμε τους ίδιους εισηγητές και συνεισηγητές. Κοιτάζω δεξιά-αριστερά για να δω ποιος από όλους αυτούς τους κυρίους είναι παρόν για να του δώσω το λόγο. Ο κύριος Σάς. Στάς. Ευχαριστώ. Είναι μια άλλη, ακόμα μια υπόθεση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που υποβάλλω αντίρρηση μαζί με τους συναδέλφους εναντίον μιας πρότασης της Κομισιόν σε αυτή την περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή κάποιων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Πρόκειται για βαμβάκι και αραβόσιτο από την AgroScience, ε, το βαμβάκι από την Bayer. Στα δύο ψηφίσματα που έχετε μπροστά σας αναφέρεται όλος ο κατάλογος των αντιρρήσεών μας. Και για το βαμβάκι και για τον αραβόσιτο. Υπάρχουν και μεμονωμένες αντιρρήσεις και κοινέ αντιρρήσεις. Καταρχά, την υπόθεση του αραβόσιτου, του βαμβακιού, συγγνώμη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει καταρχά μια θετική γνώμη τη ΕΦΣΑ, γι' αυτό ακριβώ η Κομισιόν είχε εισαγάγει αυτό το φάκελο, αλλά απέναντι σε αυτή τη θετική αξιολόγηση τη ΕΦΣΑ υπήρχε μία σειρά από επικρίσει από τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών για το βαμβάκι μεταξύ άλλων είναι ότι υπάρχουν ελλειπή στοιχεία σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση των ζυζανιοκτώνων και φυτοφαρμάκων καθώς και των καταλήπων μεταβολητών στα γενετικά τροποποιημένα φυτά και για τα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές. Επίσης για την αξιολόγηση για το περιβάλλον είχαμε λήψεις και καθώς και για το σχέδιο προστασίας του περιβάλλοντος επίσης ελλείψης, κάποιες αρχές ε, επικρίνουν ε, το γεγονός ότι βασιζόμαστε σε στοιχεία από βάσεις δεδομένων πολύ ελλειπής και ότι λάβαμε υπόψη μας πάρα πολύ λίγες έρευνες και ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη καθόλου μελέτες για την επίπτωση του βαμβακιού αυτού ε, γενετικά τροπημένου στην ανθρώπινη και ζωική υγεία. Για τον Αραβόστο υπάρχουν επικρίσεις για το ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ή γιατί λείπουν στοιχεία ή γιατί υπάρχουν εντελώς διστάμενες απόψεις. Ορισμένες ε, δοκίμες δεν έχουν γίνει, κάποια τεστ δεν έχουν ε, γίνει ποτέ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ασφάλεια είναι εντελώς, ε, αμφισβητούνται εντελώς. Υπάρχει επίσης έλλειψη στοιχείων για την τοξικότητα σε ένα κύκλο 90 ημερών. Επίσης, ε, λείπει ο πλήρης ε, διατροφικός φάκελος και για το βάμβακα και για τον αραβόσιτο. Επίσης, ε, έρευνες από ερευνητές και επιστήμονες ανεξάρτητες λένε ότι υπάρχουν ελλείψεις στις συγκριτικές μελέτες τοξικολογικής φύσεως και υπάρχουν και ανησυχίες που εκφράζονται από τους ίδιους επιστήμονες και ερευνητές για την επίπτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα αυτών των δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Στα ψηφίσματα αναφέρουμε ότι οι δύο αυτές καλλιέργειες ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δείχνουν αντοχή σε κάποια ζυζανιοκτώνα, ε, ζυζανιοκτώνα ε, το, τις γλυφοσυνικές ε, ενώσεις που θεωρούνται τοξικές και επομένως υπάρχει ένα κριτήριο εδώ πέρα ε, σε σχέση με τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα. Κανονικά ισχύει αυτός ο κανονισμός, αλλά εμείς παρεκκλίνουμε από αυτό τον κανονισμό. Επίσης, η ενεργή ουσία 2,4D δημιουργεί κίνδυνο στα έμβρια. Έχει τοξικές επιπτώσεις. Όλα αυτά τα αναφέρουμε στα ψηφίσματά μας. Είναι πολύ αρνητικές αυτές οι επιπτώσεις για την υγεία των εμβρίων. Και αν δεχτούμε τη θέση στην αγορά αυτών των οργανισμών, στην πραγματικότητα θα εξάγουμε τα προβλήματά μας προς τρίτες αγορές. Τρίτες αγορές όπου θα καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα, τρίτες χώρες που θα καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα, όπου θα αυξηθεί η χρήση ε, επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και ζυζανιοκτώνων και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει καμία συνέπεια στην πολιτική μας. Στις τρίτες χώρες δεν θα εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική προστασίας της υγείας όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα υπάρχει και ένα πρόβλημα, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εκδημοκρατικοποιηθεί. Στο μεταξύ η ομάδα μου έχει υποβάλει προτάσεις για αυτό το πρόβλημα, αλλά επίσης και οι υπόλοιποι συνεισηγητές θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το θέμα για να επιληθεί δεδομένου του προβλήματος που θέτει η διαδικασία λήψη των αποφάσεων μια και ο ίδιο ο πρόεδρο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η διαδικασία τη επιτροπολογία ουσιαστικά δεν είναι δημοκρατική, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εισαγωγή νέων ουσιών γενετικά τροποποιημένων. Είναι η 8η ή η 9η φορά που ε, παρουσιάζουμε τέτοιες αντιρρήσει πάντα με επιτυχία και στην Ολομέλεια έχουμε επιτυχία και το κάνουμε με την υποστήριξη αθρώων, ε, αθρώας πλειοψηφίας. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 128 βουλευτές που εκφράστηκαν κατά. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα συμπεράσματα που ακούσαμε στην Ολομέλεια είναι αυτά που έχουν προτεραιότητα έναντι στις μεμονωμένες φωνές που ακούγονται. Ο κύριος Παγνιό. Ε, θέλω να μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Γκυγιόν Μπαλάς που συνυπέγραψε αυτή την αντίρρηση. Καταρχάς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω από πλευράς μου κάποια πράγματα. Όλες οι αντιρρήσεις μας ε, υπεψηφίστηκαν από μια μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές οι αντιρρήσεις ε, κατατέθηκαν από εκπροσώπους έξι πολιτικών ομάδων, διαφορετικών έτσι, πολιτικών ομάδων. Αυτοί που θα ήθελαν να αμφισβητήσουν αυτές τις ε, αντιρρήσεις, να σας πω ότι αυτές οι αντιρρήσεις είναι ένα μέτρο για να εξασφαλίσουμε ότι οι επιλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται σεβαστές χάρη στα θεσμικά του προνόμια. Αυτές οι αντιρρήσεις δεν έχουν ε, να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης, το σεβασμό της ε, πλειοψηφίας των ε, βουλευτών, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική επιλογή, ούτω ώστε να αποκαταστήσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει και σέβεται τους πολίτες και πολίτησες. Πρέπει να το πούμε αυτό και κυρίως να μας ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα έχουμε δύο αντιρρήσεις μπροστά μας που αφορούν δύο ε, γενικά τροπημένους οργανισμούς ε, που είναι αντι, ε, ανθεκτικοί στα ζυζανιοκτώνα και το, ας πούμε το βαμβάκι έχει στο γλυφοσυνικό αμμόνιο ή μάλλον το γλυφοσυνικό αμμόνιο αντιστέκεται σε κάποια ζυζάνια που είναι λεπιδόπτερα. Ή επίσης υπάρχει αντίσταση στο οξύ 2,4D που προκαλεί ε, συγγενικές ανομαλίες και ε, διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα. Το αν επιτρέψουμε αυτό το, την εισαγωγή αυτού του αραβόσιτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγηθούμε σίγουρα σε μια αύξηση αυτών των καλλιεργιών στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Και επομένως θα αυξηθεί η χρήση αυτών των ζυζανιοκτώνων ε, που δεν τα θέλουμε καθόλου δηλαδή το γλυφοσυνικό αμμόνιο και το 2,4D. Αυτά λέει ο κ. Μπαλάς. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος, επιτυπεί κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί μου έχουν αναφερθεί με πολλές λεπτομέρειες ε, γιατί έχουμε καταθέσει αυτές τις ενστάσεις. Ε, μέχρι Νομίζω λοιπόν ότι ε, ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαδικασία της εξοδότησης παρουσιάζει λήψεις και εμείς θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε ενιστήσεις γιατί σας είπα η διαδικασία είναι ελλειπής και περιμένουμε ε, την έρευνα να επιβεβαιώσει τα βασικά κενά που υπάρχουν ε, στην, ε, στις έρευνες τις τοξικολογικές, τις επιπτώσεις ενδεχομένως στο ανοσιοποιητικό σύστημα. Ο δικός μας ο στόχος είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η αρχή της πρόληψης και όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι ισχύει το μέγιστο επίπεδο προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να αγνοεί αυτές τις, ε, ε, την κριτική που προέρχεται από τα κράτη-μέλη ε, δεν υπάρχουν ε, ε, ικανοποιητικές δοκιμές. Εμείς λοιπόν είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε μια λύση. Αλλά μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμεθα και να καταθέτουμε ένσταση για μια ελλειπή διαδικασία εξου... μάλλον. Αδειοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε παρεμβαίνω εξ του ΕΛΚ και εμείς θα ακολουθήσουμε το ίδιο κριτήριο. Πρόκειται για δύο προϊόντα που έχουν τύχει αδειοδότησης, όχι για καλλιέργεια βεβαίως, πρόκειται για μία εκτελεστική ε, πράξη και τίθενται δύο ερωτήματα. Εάν η Επιτροπή ακολούθησε την εντολή της ή όχι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κακή χρήση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν υπάρχουν ε, επιστημονικές αξιολογήσεις, θα πρέπει να τις έχουμε. Να αναλύσουμε δηλαδή τους ενδεχόμενους ε, κινδύνους και αν έχουν γίνει οι κατάλληλες αξιολογήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις περιπτώσεις ε, υπάρχει θετική γνωμοδότηση και για το συγκεκριμένο βαμβάκι και τον, ε, και τον αραβόσιτο. Σε σχέση με τη ζημία που θα μπορούσαν, τη βλάβη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στην ανθρώπινη υγεία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν πρόκειται για σπόρους, για καλλιέργεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε αυτές τις αντιρρήσεις, διότι στο Συμβούλιο διαμορφώθηκε μία θετική άποψη και νομίζω ότι οι αντιρρήσεις αυτές προβάλλονται για λόγους κινητοποίησης της κοινή γνώμης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν και προηγουμένω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα διέξοδο στην ε, έγκριση των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ε, πρέπει λοιπόν να αρτεί αυτό το αδιέξοδο και να μην χρησιμοποιούμε τις εγκρίσεις ως μια δικαιολογία. Πρέπει να ε, ακολουθήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Εμεί δεν είμαστε επιστήμονες, είμαστε πολιτικοί και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις ε, που να μην είναι τεκμηριωμένες. Βασιζόμαστε στα στοιχεία τα οποία μας δίδει η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ. Δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Αν όχι, από την Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε και δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εξηγήσει το σκεπτικό των ε, προτάσεων. Εγώ θέλω να φέρω πέντε ε, στοιχεία. Πρώτον, η αναφορά για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς γενικά, αλλά και για το βαμβάκι ειδικότερα, όλα αυτά βασίζονται αυστηρά στην ε, νομοθεσία. Κατόπιν η ΕΦΣΑ θα πρέπει να έχει προβεί σε αξιολόγηση κινδύνων και για τα δύο προϊόντα. Θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσει στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς κατά νου ότι τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν την αξιολόγηση κινδύνων. Και η ΕΦΣΑ έχει επίσης σχολιάσει και τα σχόλια της ΕΦΣΑ. Ε, εξάλλου και η κοινή γνώμη είχε την ευκαιρία και αυτή να σχολιάσει και η ΕΦΣΑ έχει και αυτή σχολιάσει τα σχόλια του κοινού. Ε, το πέμπτο σημείο είναι ότι τα σχέδια των αποφάσεων συμβαδίζουν με το στόχο του κανονισμού που είναι να προστατεύει τη υγεία των ανθρώπων, των ζώων και το περιβάλλον. Κατόπιν τούτου, οι αποφάσεις ε, ψηφίστηκαν στις 27 Μαρτίου στη Μόνιμη Επιτροπή χωρίς ε, γνωμοδότηση. Είναι όμως πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι λόγοι για το ότι τα κράτη-μέλη δεν τοποθετήθηκαν, ούτε καταψήφισαν, ούτε δήλωσαν στην αποχή, Οι λόγοι είναι πολιτικοί και διότι υπάρχει αρνητική άποψη στην κοινή γνώμη. Ως εκ τούτου αναμφίβολα έχουμε παραμείνει πιστοί στις διαδικασίες ε, και θέλω να υπογραμμίσω ότι ε, το Κοινοβούλιο έχει περισμένο δικαίωμα ελέγχου, δηλαδή ε, κατά πόσον ισχύει αυτό στον, στον, στην εφαρμοστική πράξη. Εμείς ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχόλια και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ δύο σχόλια. Όσον αφορά τα ε, φυτοφάρμακα, όπως είπε και η κυρία Αγιούζο, ε, υπάρχει σχετική νομοθεσία περί φυτοφαρμάκων. Καταρχήν, αυτά τα δύο προϊόντα θα προβλέπονται για εισαγωγή. Άρα, δηλαδή, αν υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει στο περιβάλλον, αυτέ θα υπάρχουν ε, σε τρίτη χώρα και όχι στην Ευρώπη. Δεύτερον, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι τα κατάλοιπα ή η νομοθεσία για τα παρασιτοκτόνα ε, βασίζεται και ισχύει για όλες τις αγωγές είτε είναι για μεταλλαγμένα προϊόντα είτε όχι. Ως εκ τούτου και αυτά ε, θα πρέπει να καλύπτουν τις ε, πολύ υψηλέ προδιαγραφές για τα παρασιτοκτόνα. Τώρα έχουν κατευθεί δύο προτάσεις. Επί της ε, πρώτης, δυστυχώ το Κοινοβούλιο καταψήφισε, είναι η πρώτη εκείνη που δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να απορρίπτουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς εφόσον υπάρχουν ε, αποχρόντες λόγοι. Αυτό συνέβη και θέλουμε να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις με το Συμβούλιο. Ε, όπως αναφέρθηκε και από έναν κύριο Ευρωβουλευτή, ο πρόεδρος κ. Γιούγκερ πρότεινε άλλο ένα μέτρο για να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία της επιτροπολογίας. Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι μέχρι να εγκριθεί αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που ισχύουν, γιατί αν δεν το κάνουμε ε, τότε προφανώς προφανώς ε, θα βρεθούμε σε δυσκολία. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι εμείς ακολουθήσαμε τις διαδικασίες ότι δεν ξεπεράσαμε τις εφαρμοστικές μας αρμοδιότητες και ως εκ τούτου δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να αποσύρουμε την πρόταση. Κατά τα άλλα, ε, πρόκειται να υπάρξει ψηφοφορία στις 16 Μαΐου. Νομίζω λοιπόν αυτά που σας είπα, οι εξηγήσει που έδωσα, να εξηγούν και τη θέση της Επιτροπής. Επίσης, ελπίζω να κατέστη σαφής υποχρεωσή μας, δηλαδή στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ να υπενθυμίσω στους ε, συναδέλφους ότι από αυτή τη ε, αντίρρηση θα ψηφίσουμε αύριο. Η τρίτη αντίρρηση με βάση τον κανόνα 106 αφορά στα συμπεράσματα LCP η κυρία Κονέτσνα. Ε, μόλις την είδα να μπαίνει στην αίθουσα, παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Γνωρίζω ότι ο υδράργυρος και τα οξύδια του αζότου έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Γι' αυτό ήθελα να μειώσουμε τις ε, εθνικές ε, προδιαγραφές και ανώτατα όρια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει η πρόταση της Επιτροπής να γίνει πιο αυστηρή, αλλά δεν ε, ήταν επαρκής. Αυτή τη στιγμή η οδηγία βρίσκεται σε τριμερή διάλογο και πιστεύω ότι η μείωση των εκπομπών θα πρέπει να συμβαδίζει με ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο και αυτό θα πρέπει να, τονίζουμε, να το τονίζουμε κάθε φορά όταν η Επιτροπή υπερβαίνει τα ε, όρια, της, τα όρια που θα έπρεπε. Όπως ισχύει στην περίπτωση του λιγνίτη των οξυδίων του αζότου και του ε, υδράργυρου. Η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση δημοσιοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, αυτά τα BATs, που είναι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν με βάση τις τεχνολογίες εχμής και τα πλεονεκτήματα ζητήματα που ενέχουν πέρα από το κατά πόσο αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε λοιπόν τεχνικές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δεν ε, ελήφθησαν υπόψη οι σωστές προδιαγραφές και η Επιτροπή δεν αντέδρασε. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να ε, φτάσουμε στην αντιμετώπιση του κινδύνου σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς τα συμπεράσματα των BAT ο ε, οδήγησαν σε λάθη από την Επιτροπή. Δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου του 2016 η Επιτροπή δεν επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν τις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Άρα τα αποτελέσματα δεν ήταν σωστά. Ως ε, προς το υδράργυρο και την καύση του λιγνίτη, τα στοιχεία των BATs ήταν εν μέρη λανθασμένα, γιατί δεν έγιναν επαληθεύσεις από το EIBCB ιδιαίτερα σε σχέση με την, τα όρια που ισχύουν σε επίπεδο ΙΠΑ. Και γι' αυτό δεν, δεν ελήφθησαν υπόψη τα όρια όπως είχαν προοριστεί. Γι' αυτό και δεν υπάρχει το, ε, τα όρια, δεν υπάρχουν τα όρια όπως ορίζονται από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Η διαδικασία της βέλτης της διαθέσιμης τεχνολογίας των BAT ε, ε, αφορούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει καύση λιγνίτη ε, που να καίγεται όπως θα έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι στην Τσεχία υπάρχει καύση άνθρακα και αυτή είναι η μόνη πηγή θέρμανσης που υπάρχει και υπάρχουν ολέθριες συνέπειες για το ενεργειακό ε, μείγμα. Σε σχέση με το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος ορίζει το δικό του BAT σε σχέση με την αποθήκευση των καυσίμων. Γι' αυτό ίσως έχουμε να κάνουμε με παραβίαση των συνθήκων. Δυστυχώς, τα 28 Απριλίου, τα κράτη-μέλη αποφάνθηκαν επί των BATs χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Και όλα τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να μην χρησιμοποιούν το λιγνίτι στο ενεργειακό τους μείγμα εκτός από την Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ειδική κατάσταση της Ελλάδας γιατί μιλάμε και για τον ισιωτικό της χαρακτήρα. Άρα η απόφαση για τη ε, βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία δεν ήταν ε, σωστή γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο λιγνίτης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια του ενεργειακού μείγματος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεροληψία σε σχέση με τη χρήση του λιγνίτη. Για το BAT υπέρ τάχθηκε η Γερμανία η οποία υποστηρίζει τις ανανεώσιμες και τα συμπεράσματα BAT θα πρέπει να ισχύουν τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα και αυτή, σε αυτή την περίπτωση ούτε η Γερμανία δεν μπορεί να ε, λειτουργήσει χωρίς μονάδες λιγνίτη. Πόσο μάλλον η Τσεχία ή η Βουλγαρία. Λυπάμαι διότι η Επιτροπή επέτρεψε κάτι τέτοιο και δεν προέβαλε τη σωστή επιχειρηματολογή. Ε, πολλοί το θεωρούν νίκη μέσα στα πλαίσια της επιτροπολογίας, αλλά αυτές οι νίκες ε, μάλλον πλήττουν όλους τους υπόλοιπους σε σχέση με την ε, εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη. Έχουμε ένα πολιτικοποιημένο κείμενο. Μπορεί να θεωρείτε ότι δεν αφορά τη χώρα σας γιατί δεν χρησιμοποιείτε λιγνίτη, αλλά σήμερα είναι ο λιγνίτης, αύριο μπορεί να είναι κάτι, κάτι άλλο. Γι' αυτό προβάλλουμε αυτή την αντίρρηση. Λοιπόν, ε, η Σκιώδηστο, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως εξήγησε και η κυρία Κονέτσνα, το να μιλάμε για τον λιγνίτη και τις εγκαταστάσεις κάψης με λιγνίτη, ε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι ε, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις εκπομπές, να φτάσουν οι εκπομπές αυτές σε μηδενική βάση στο μέλλον. Ε, εδώ μιλάμε για την ε, μη εφαρμοστική πράξη η οποία σχετίζεται με μια οδηγία του 2010. Ε, τώρα είμαστε στο 2017. Θα ήθελα λοιπόν να δράξω αυτή την ευκαιρία επειδή ψηφίζουμε αύριο για να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν, πόσες, για, πώς, για ποιες βιομηχανικές μονάδες μιλάμε. Μιλάμε για δεκάδες ε, χιλιάδες. Όταν ε, μιλάμε για μονάδες καύσης με λιγνίτη, μιλάμε για εκατοντάδες, για χιλιάδες. Ε, δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό, διότι όπως σας είπα, Μιλάμε για μια οδηγία του 2010, μιλάμε για δεδομένα του 2010, είμαστε 7 χρόνια αργότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εντωμεταξύ έχει ε, προκύψει και νέα τεχνολογία. Αυτό που επίσης ε, ενδιαφέρει είναι ότι μιλάμε για το Μιλάμε για οξύδια του αζότου, αλλά ε, πρέπει να έχουμε υπόψη και κάποιες κατά νου και κάποιες διαφορές. Ε, πρακτικά, τι σημαίνουν όλα αυτά. Οι αρμόδιες αρχές ε, πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ε, τώρα, όσον αφορά το κόστος, γιατί έγινε λόγος και για το κόστος, κυρίως στις παλαιότερες εγκαταστάσεις, το κόστος που θα προκύψει για αυτές τις εγκαταστάσεις ε, το κόστος αυτό θα είναι δυσανάλογο. Ε, τι σημαίνει αυτό στην πρακτική, δηλαδή θα αξιολογείται ε, κατά περίπτωση ή θα υπάρχει μια γενική απόφαση. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, οι Πολωνοί συνάδελφοι επίσης αναφέρθηκαν και στην δυνατότητα ή στο φόβο περισσότερο του να υπάρξει blackout. Blackout κατά διάρκεια διαφόρων εργασιών ε, ε, επιδιόρθωσης και επισκευής. Ένα τέτοιο blackout ε, είναι σοβαρή υπόθεση. Πρέπει πραγματικά να το λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχει τέτοιο κίνδυνο Και ποιο θα ήταν, τι θα σήμαινε αυτό για την κοινωνία. ίσως μπορώ να κάνω και κάποιες άλλες εμπληρωματικές ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε, γιατί όλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα για να δούμε πώς θα ψηφίσουμε αύριο. Πρόεδρος, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 5 ώρα θα έρθει ο Επίτροπος για να μιλήσουμε για το διαρθρωτικό διάλογο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να είσαστε σύντομοι στα σχόλιά σας για αυτή την αντίρρηση, όσο πιο σύντομοι γίνεται βέβαια. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ντάνς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Μιλάμε για περίπου 500.000 άνθρωποι που πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο Επίσης υπάρχει και άλλος ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που πεθαίνουν λόγω των εκπομπών των μονάδων με καύση τον άνθρακα, με καύσιμο υλικό τον άνθρακα. Το θέμα είναι ότι αυτά που είπε η κυρία να φοβάμαι ότι δεν ισχύουν, δεν είναι αλήθεια. Είπε ότι δεν υπάρχουν ε, κάποιες μονάδες ε, λιγνίτη που να καλύπτουν τα όρια. Υπάρχουν. Υπάρχουν αυτές που καλύπτουν τα 750 mg, Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ε, δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές. Και πάρα πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε εδώ είναι του 2010. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, πάρα πολλές μονάδες ε, καλύπτουν τα όρια που έχουν καθοριστεί με το ίμιση της υπάρχουσας ε, τεχνολογίας. Πολλές από αυτές τις ε, μονάδες έχουν κατασκευαστεί το 1975, άρα δηλαδή είναι δυνατόν να μειωθούν εκπομπές από μονάδες που χρησιμοποιούν λιγνίτη, να μειωθούν περαιτέρω εκπομπές. Και τα μέτρα που εξετάζουμε εδώ με τη διαδικασία των βέλτιστων τεχνικών, των βέλτιστων διαθέσιμων, της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, αυτά έχουν στόχο το να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση. Δηλαδή, όταν ε, δεν θα υπάρχει αυτή η τεχνολογία, ο λιγνίτης ε, είναι ε, ο λιγότερο, το λιγότερο ρηπαίνον κάψιμο. Και αυτό είναι γεγονός. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την απαραίτητη τεχνολογία, γιατί υπάρχει αυτή η τεχνολογία και εκείνο με το οποίο εμείς διαφωνούμε, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αντίρρηση, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβαστικές ε, προτάσει και αυτές όμως προχωράνε πάρα πολύ και δεν αφορούν μόνο τη γνώση που υπάρχει για την τεχνολογία, αλλά αφορούν και τη συμπερίληψη της βιομηχανίας στις συζητήσεις για να επιτευχθεί συμβιβασμό. Και επειδή δεν υπάρχει ε, συμβιβασμό, ε, δεν έχουμε επιτύχει και την βέλτιστη δυνατή μείωση. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το κατά πόσον υπάρχουν πολλές μονάδες ε, οι οποίες προσπαθούν να μειώσουν τις ε, εκπομπές ε, που έχουν επενδύσει δηλαδή σε αυτήν την τεχνολογία. Εγώ νομίζω ότι ε, θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά αυτέ οι βιομηχανικέ μονάδε, οι οποίε έχουν καταβάλει μεγάλε προσπάθειε για να μειώσουν τι εκπομπέ. Γνωρίζουμε παραδείγματο χάρη ότι οι φτωχότεροι στην κοινωνία μα υποφέρουν περισσότερο από τη μόλυνση ρήπανση του αέρα. Ε, πολλοί θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται ακριβώ σε αυτή τη ρήπανση τη ατμόσφαιρας και είναι ένα τεράστιο κόστο για το σύστημα υγεία των κρατών μελών μας. Ε, είναι λοιπόν πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι ασθένειες που προκύπτουν ακριβώς λόγω της, ε, της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την αντίρρηση γιατί πετάει στα σκουπίδια αυτές τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει να διασωθεί η ζωή πολλών ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει καλή σημαντική δουλειά και θα ήταν λάθος και ανοησία να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Κύριε Βυζνιεύσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κονέτσινα για την εκτελεστική πράξη, η οποία θέλει να μας εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες για τα εργοστάσια που και είναι λιγνίτη. ούτως ώστε να έχουμε ω να πιο χαμελές εκπομπέ οξυδίων του αζότου. 175 ε, μιλιγκράμμ για τα οξύδια του αζότου. Αυτό είναι το σχέδιο. Συνήθω είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές τις ε, μονάδες ε, λόγω της γεωλογική και γεωγραφική του κατάσταση. Αυτοί που συμφώνησαν ε, κλείνουν τα μάτια σε δύο πράγματα. Καταρχάς, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπομπών οξυδίου του οξυδίων του αζότου προέρχονται από τις μεταφορές και όχι από τις μονάδες ε, που καίνε λιγνίτη. Ε, τα όρια που βάζουμε για τις ε, μονάδες αυτές του λιγνίτη δεν θα επιτρέψουν να λύσουμε το πρόβλημα και να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, αλλά αυτό θα ε, επηρεάσει την ε, τιμή της ενέργειας και την ε, διαθεσιμότητα της ενέργειας. Δεύτερον, αυτή η οδηγία λέει ξεκάθαρα ότι η οικονομική απόδοση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τη στιγμή που αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές τεχνικές. Αλλά αυτό όμως δεν ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν. Ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι για τις μεγάλες εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε παρεκκλήσεις. Και τα όργανα, ε, οι φορείς που παίρνουν αποφάσεις, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το χρόνο που χρειάζονται αυτές οι εγκαταστάσεις για να εξυγχρονιστούν. Στο μεταξύ θα πρέπει όμως να μην να ξεμείνουμε από ενέργεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια. Μία ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να λάβει υπόψη και το κόστος μη παραγωγής ενέργειας κατά την περίοδο αυτή που θα γίνονται εργασίες για να εξυγχρονιστούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Το να φτάσουμε σε, στα όρια 175 μιλιγκράμμ για τα οξύδια του αζότου θα, έχουν, θα, θα έχει σαν συνέπεια ότι για τις εγκαταστάσεις που συχνά είναι στα όρια της βιωσιμότητας θα πρέπει να γίνουν ε, πάρα πολύ δαπανηρές ε, ε επενδύσεις που δεν έχουν κανένα οικονομικά για να εξυγχρονιστούν. Και θα έχουν πολύ περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον. Αυτό είναι μια απειλή. Κινδυνεύουν αυτά τα εργοστάσια να κλείσουν πριν την ώρα τους ή να μην μπορέσουν να παράγουν ενέργεια. Και μπορεί στην Πολωνία σε λίγα χρόνια να μην έχουμε πια δυνατότητα, επαρκή δυνατότητα παραγωγής για να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών. Θα φτάναμε στην παράλογη κατάσταση, όπου τα, κράτη τα οποία δεν χρησιμοποιούν το κάρβουνο ή το λιγνίτη, μαζί με την Κομισιόν υποδεικνύουν στα υπόλοιπα κράτη τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα καύσιμα υλικά, τι πρέπει να κάνουν. Και τους λένε ότι δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσετε αυτέ τι πρώτε ύλες ε, λέγοντάς μας ότι δεν έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Όμω πρέπει να ξέρετε, τα 10 τελευταία χρόνια μειώσαμε τι εκπομπέ στην Πολωνία ε, εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου, ειδικά από τι εγκαταστάσει αυτέ παραγωγή ενέργεια κατά 50%. Και για τα οξύδια του αζότου έχουμε μία μείωση των εκπομπών οξυδίου του αζότου κατά 20%. Οι τεχνολογικές όμως ε, πρόοδοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Πάντα έχουν όρια, έχουν τα όρια τους. Σήμερα θα πρέπει να κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να έχουμε ελάχιστη ε, πρόοδο. Και το κόστος αυτής της πρόοδου θα μπορούσε να είναι μία αύξηση της ενεργειακής στόχιας στις χώρες όπου η ενέργεια βασίζεται στο κάρβουνο και στο λιγνίτη. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλουν τα άτομα τα οποία συνέταξαν αυτό το κείμενο. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ρεαλιστικούς στόχους, ε, χωρίς να ξεχνάτε και ε, το καλό του πολίτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι. Αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Υπάρχουν κάποια λάθος στοιχεία ε, που αναφέρονται σε αυτό το ψήφισμα. Είμαι λιγάκι απογοητευμένος που, γράφ, που διαβάζοντας αυτή την αντίρρηση, γιατί νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που γράφουμε είναι σωστό. Να μην έχει λάθος στοιχεία. Πρέπει να πω ξεκάθαρα από την αρχή ότι δεν είμαι ικανοποιημένο ε, με το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαφή συμβιβασμό. Φυσικά θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ πιο αυστηρά πρότυπα. Αυτή ήταν μια διαδικασία εξαετή. Έξι χρόνια μα πήρε. Αν τελικά στο ψήφισμα ε, αναφερθούμε μόνο σε μια συνάντηση τον Οκτώβριο του 2016, ξέροντα ότι αυτή είναι μια διαδικασία εξαετή, στην πραγματικότητα βασιζόμαστε ε, και αν βάλουμε τα πρότυπά μας ε, σε αυτά που ξέραμε το 2010 είναι λάθος. Τώρα ξέρουμε που μπορεί να πάει ο κλάδος και ο τομέας αυτός. Τέλο πάντων, είναι πολιτικός συμβασμός αλλά στην πραγματικότητα αγναγνωρίζεται, τα, παραγνωρίζεται τα στοιχεία. Για τον υδράργυρο, εμείς είπαμε ότι τα επίπεδα θα πρέπει να μειωθούν, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πηγή. Αν διαβάσετε όμως τις πληροφορίες που υπάρχουν στην οδηγία, 80% των εγκαταστάσεων λιγνίτη πληρούν τα πρότυπα τα οποία έχουν ε, ήδη τεθεί ε, για το 2021 και τα πληρούν σήμερα. Τι είναι το, το αδύνατο δηλαδή. Για τα οξύδια του αζότου ε, αναφέρεται ε, το ETS. Το ETS όμως δεν αναφέρεται στα οξύδια του αζότου γιατί δεν είναι αέριο του θερμοκηπίου. Εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το κείμενο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και ξέρετε ότι πολλές εγκαταστάσεις λιγνίτη σέβονται αυτά τα όρια τα οποία έχουν τεθεί εδώ μόνο με πρωτογενή μέτρα. Μετά το 2010 είχαμε νέες μετρήσεις και νέα μέτρα τα οποία μας ε, επιτρέπουν να προβούμε σε περαιτέρω ε, μειώσεις και για τον υδράργιο ε, μπορούμε να σεβαστούμε τα όρια. Υπάρχουν βέβαια διάφορες παρεκκλήσεις εντός του κειμένου. Εάν πούμε ότι έχουμε αντίρρηση γιατί αυτό είναι πολύ αδύναμο, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά εάν το πάμε αντίθετα, στην πραγματικότητα το ψήφισμα αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Είναι πολύ λάθος και γι' αυτό συνιστώ θερμά στους ε, συναδέλφους να μην υποστηρίξουν αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα σήμερα. Το σημείο εκκίνησης είναι ότι την Παρασκευή, ε, την Παρασκευή 28 του μηνός ενέκρινε η Επιτροπή αυτό το πλαίσιο και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, μελλοντικές προκλήσεις ως προς την ποιότητα του αέρα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το θέμα των πρόωρων θανάτων των 400.000 είναι κάτι που μας απασχολεί. Ας δούμε όμως ε, πώς είχε η συζήτηση των LCP. Οι εγκαταστάσεις λιγνίτη, μιλάμε για 18% ε, οξυδίων του αζότου και 19% υδραργύρου. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει άμεση ε, συνδεσιμότητα με την οδηγία και με την ποιότητα του αέρα. Υπάρχει μία πολύ σοβαρή παραβίαση. Έχουμε 16 παραβιάσεις σε σχέση με τα οξύδια του αζότου και τα οξύδια του θείου. Η κατάσταση λοιπόν είναι πραγματικά πολύ δυσίωνη. Όταν μιλάμε για την ίδια τη διαδικασία ε, υπήρξαν πολλοί ισχυρισμοί, σοβαροί ισχυρισμοί για το κατά πόσα ήταν εύρωστη όλη η διαδικασία που ακολουθήσαμε. Ε, και ε, θα ήθελα να πω ότι για τις εγκαταστάσεις λιγνίτη και το BAT είχαμε διεξοδικές μελέτες τα τελευταία έξι χρόνια μετά από σύσταση της ε, Επιτροπής. Είχαμε το 12ο μπρεφ και αυτή η διαδικασία έχει δοκιμαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, δηλαδή εξάγουμε αυτή την πλαισίωση μελέτης χάρη στην ποιότητά της. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μία ε, εις βάθος ανάλυση και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα δεδομένα. Μιλάμε για μία ομάδα 289 μελών που περιλαμβάνει όλους τους ε, τομείς ε, με ολόκληρο, με όλους τους τομείς ε, δηλαδή της βιομηχανίας, ακαδημαϊκούς και κοινωνία των πολιτών. Το 2011 συστάθηκε η Επιτροπή και ολοκλήρωσε τις εργασίες το 2016. Ε, κάλυψε στοιχεία από 580 ομάδες και 220 μελέτες, καθώς και 8.100 σχόλια τα οποία ε, δημοσιεύτηκαν στην τελευταία συνάντηση της τεχνικής ομάδας είχαμε όλα τα στοιχεία BAT, ε, δηλαδή της βέλτιστης διαθέσιμης ε, τεχνολογίας. Είχαμε 140 επιρογνώμονες για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Ελπίζω αυτά τα στοιχεία να δείχνουν πόσο σοβαρή είναι αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ σοβαρή λόγω ε, διεξοδικής μελέτης μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας BAT, της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το BAT-AL γιατί καλύψαμε όλους τους τομείς, επτά δηλαδή στο σύνολο. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν 74 συμπεράσματα. Τα 72 αφορούν ε, την αποτελεσματικότητα, 15 BAT και 270 ε, συμπεράσματα για την ποιότητα του αέρα. Είναι πολύ αυστηρή διαδικασία και δεν μπορείτε να μιλάτε για πολιτικοποιημένη διαδικασία. Είναι η πιο αυστηρή δυνατή και νομίζω ότι ε, τιμούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ακούσαμε επικρίσεις από ΜΚΙΟ αλλά και από την Επιτροπή ότι δηλαδή τα έγγραφα αναφοράς ε, βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ακολούθησαν την διαδικασία πίεσης και λόμπινγκ από την ε, βιομηχανία. ή ότι έγινε λόμπινγκ με τις ΜΚΟ. Μα αν έγινε κάτι τέτοιο τότε ακολουθήσαμε όλο το φάσμα. Και στο τέλος ο Ευρωπαίος πολίτης αμείβεται από αυτή τη διαδικασία γιατί μιλήσαμε για 400.000 θανάτους από την κακή ποιότητα του αέρα και κατανοείτε ότι αυτή είναι μία πολύ θετική διαδικασία. Οι αντιρρήσεις μας είναι γνωστές, τις ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ένα ειδικό λόμπι ε, μας πίεσε, δηλαδή η Euracall. Νομίζω ότι υπάρχει ένα εμπλεκόμενο, ένα ενεχόμενο κόστος, το οποίο δεν αποκρύψαμε θέλουμε να μειώσουμε τις δαπάνες γιατί δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη διαδικασία. Όμως η διαδικασία είναι εύρωστη και φτάνει σε απτά συμπεράσματα και δεν θα πρέπει να δούμε μόνο το βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά και τα ευεργετήματα σε σχέση με τις καινοτομίες και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και λαμβάνουμε υπόψη και συνιστώσεις, τις συνιστώσεις υγείας που είναι στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Άρα πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία που είναι πολύ σημαντική για μας γιατί το να λέτε ότι οι συμμετέχοντες δεν εξέφρασαν την άποψή τους το 2006 ή να επικρίνεται... Ε, τα συμπεράσματα για το λιγνίτι και τον υδράργυρο είναι κάτι το απαράδεκτο. Νομίζω ότι σας έδωσα στοιχεία για το μη βάσιμο των επικρίσεων σε σχέση με το ε, EIPCB. Η διαδικασία είναι παραδειγματική και αυτό το αναφέρω για άλλη μία φορά. Με συγχωρείτε, πρέπει να σας διακόψω, λέει η Πρόεδρος γιατί έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Θέλω να έχετε όλα τα στοιχεία επιτάπητος. Τρία σημεία λοιπόν. Ως προς τον τύπο στις 20 Οκτωβρίου αποφασίσαμε το φόρουμ αυτό δεν αποτελεί συνέχεια της τεχνικής ομάδας. τεχνική εργασία έχει λήξει στο έγγραφο της Μπρεφ, όχι πρέπει να επιμείνω, λέει η Πρόεδρος. Δεν, δεν γίνεται, δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση για το φόρουμ. Το φόρουμ θέλει να προβεί στην ε, ταξινόμηση των απόψεων και αυτό το τονίσαμε και κατά τις συζητήσεις οι οποίες ήταν εκτενείς, γιατί θέλαμε όλες οι απόψεις να εισακουστούν. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Ως προς τον υδράργυρο τώρα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε κάθε ανθρωπογενή εκπομπή υδραργύρου. Και αυτό έγινε με τη νέα οδηγία για τον υδράργυρο. Και όπως ξέρετε θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του λιγνίτη. Προτείναμε λοιπόν ε, στο BAT να λάβουμε υπόψη όλες τις ε, μονάδες και να δούμε το ένα μικρογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτό είναι το κάτω άκρο γιατί ξέρετε ότι η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία αφορά τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Και η αντίρρηση βασίζεται σε παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα για το κατώτατο και ανώτατο όριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε θα έχετε και άλλη ευκαιρία να μπείτε σε λεπτομέρεια. Η κυρία Κονέτσνα μόνο για ένα λεπτό. Αν όχι, ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε αύριο και τώρα θα καλέσουμε τον Επίτροπο τον κύριο Ανδριουκάητης. Καλησπέρα, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στα πλαίσια του διαρθωμένου διαλόγου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το πεδίο της αρμοδιότητάς σας. Οι συνάδελφοι, φαντάζομαι, θα θέλουν να θέσουν τα θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου. Δεν θα πω πολλά. Ε, σας καλωσορίζω απλώς. Θέλω να, να ακούσω τις προτεραιότητες που έχετε ως Επίτροπος για τα επόμενα χρόνια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να καθίσω εδώ, από αυτή την πλευρά, λόγω του προβλήματος που έχω. Σας ευχαριστώ που επιτρέπετε αυτή την εξαίρεση. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, με μεγάλη χαρά επανέρχομαι για τον τρίτο διαρθρωμένο διάλογο ε, στα πλαίσια της, ε, Επιτροπή της Επιτροπής αυτής το 2017. Ως Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια θα ήθελα να τονίσω εν συντομία ε, λίγα σημεία που είναι του χαρτοφυλακίου μου, της αρμοδιότητάς μου. Ε, έχω πει κατ' επανάληψη το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, η προστασία, η, πρόθεση, η προώθηση και η συμμετοχή. Η υγεία θα πρέπει να ιδωθεί υπό αυτό το πρίσμα. Ε, θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ένα, μια κατάσταση πλήρους κοινωνικής, φυσικής και πνευματικής κατάστασης. Ε, πιστεύω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να είναι πιο δραστήριες για να προλάβουν και να προωθήσουν την ε, δημόσια υγεία με βάση διάφορα εργαλεία. Θα πρέπει αυτά τα μέτρα να αφορούν όλους και τους πιο ευάλωτους τους ε, φτωχούς, τους ε, άνεργους, τους ανασφάλιστους, ε, τους, τις μειονότητες όπως τους Ρωμά, να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί λόγοι, οι συμπεριφερειολογικοί λόγοι κτλ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές για να προωθήσουν την υγεία και να προλάβουν ε, και να διαχειριστούν τις χρόνιες αρρώστιες και θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες ε, τεχνικές. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Καταρχάς, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από διαφημίσεις που, για, τα, για το αλκοόλ, ας πούμε, ή για τα τσιγάρα. Επίση, η οδηγία για τον οπτικοακουστικό τομέα εδώ ε, συζητάει αυτά τα θέματα. Επίση, η οδηγία για την προστασία από τον καπνό ε, προάγει μια σειρά από project για τη μείωση των ε, λοιπόν των ζαχάρων και των λιπαρών τρανς για την διατροφή. Θα γίνει μια αξιολόγηση του κανονισμού για την, τους ισχυρισμούς για την υγεία ε, και για τη διατροφική αξία, θα πρέπει όσοι θέλουν να τονίσουν τις θετικές ιδιότητες των προϊόντων τους ε, να σέβονται ε, κάποιες, κάποιους κανόνες. Θα γίνει αξιολόγηση τέλος του 18, και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 18. θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να φέρετε το διατροφικό προφίλ. είναι ε, βασικό στοιχείο της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωση. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τους κατασκευαστές τροφίμων και τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε την ε, θρεπτική αξία των τροφίμων που είναι επεξεργασμένα. Ε, επίσης υπάρχουν πρωτοβουλίε από τα κράτη-μέλη για αυτά τα θέματα, με συγκεκριμένα βήματα για να υποστρίξουμε τι εθνικέ δράσει. επίσης, Υπάρχουν διάφορε δεσμεύσει σε αυτόν τον τομέα. Ένα ε, τομέα ε, σημασία είναι ότι τα συστατικά και οι, οι ετικέτε των αλκοολούχων ποτών. Ε, έχουμε μία έκθεση που υιοθετήσαμε 13 Μαρτίου. καλέσαμε τον κλάδο να αναπτύξει μέσα σε ένα χρόνο μία πρόταση ούτω ώστε να δίνει πληροφορίε για συστατικά και την θρεπτική αξία όλων των αλκοολούχων ποτών. Αν όμως ε, δεν ε, καλύψουμε τις προσδοκίες, θα ξεκινήσουμε μία μελέτη αντικτύπου ε, για να δούμε και τι άλλες επιλογές έχουμε. συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ανησυχώ ιδιαιτέρως για τα εμβόλια. Είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα άτομα στην Ευρώπη να πεθαίνουν ακόμα από αρρώστιες όπως η, λαρά που μπορούν να προληφθούν μέσω εμβολίων εύκολα. 500.000 άτομα ε, έπαθαν ε, η λαρά τους τελευταίους τέσσερις μήνες και διάφοροι πέθαναν. Γι' αυτό ακριβώς ε, προωθούμε μία κοινή δράση για να υποστηρίσουμε την ε, δράση των κρατών μελών για τα εμβόλια έχω συγκαλέσει ένα εργαστήρι με όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητήσουμε πώς θα βελτιώσουμε τα προγράμματα εμβολιασμού και διάδοσής τους. Σας ενθαρρύνω να είσαστε πολύ δραστήριοι για αυτό το θέμα, να το, δια, διαφημίσετε. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ε, καταπολεμήσουμε την, τον δισταγμό που υπάρχει απέναντι στα εμβόλια στην Ευρώπη. Και τώρα ας πάω στη μικροβιακή αντοχή. Ε, είναι ένας από τους πυλώνες του ε, χαρτοφυλακίου μου. Μία πρόσφατη ε, ε, αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 2011-2016 σημείωσε σημαντικές πρόοδους, αλλά κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε την μικροβιακή αντοχή με πιο συντονισμένο τρόπο. Ένα νέο ενισχυμένο σχέδιο δράσης θα προωθηθεί αργότερα μέσα στο 2017 με τρεις στρατηγικούς πυλώνες. Καταρχάς, να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία, να υπάρξει μια διεθνής, ε, ε, ισχυρή διεθνή ουσία για να συνδιαμορφώσουμε τις ε, διεθνεί δραστηριότητε και να γίνει η Ευρώπη η περιοχή με τι καλύτερε πρακτικέ. Ε, επίσης θα παρουσιάσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ανθρώπινη ιατρική. Θα σας καλώ επίσης να ζητήσετε το Συμβούλιο να επιταχύνει τη δουλειά για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τα, τις ζωοτροφές με φάρμακα που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση μικροβιακής αντοχής. Ας πάμε τώρα στα φυτοφάρμακα. Ε, το συζητήσατε στο Μάρτιο στην Ολομέλεια. Ο στόχος της Κομισιόν είναι να ενισχύσει την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία, να ενισχύσουμε τις ε, αρμόδιες αρχές για να δουν εάν νέα ε, μια νέα παρέμβαση, παραδείγματο χάρη στα φαρμακευτικά, μπορεί να αποτελεί ε, σημαντική προσθέμενη αξία. Οι υπηρεσίε μου αναλύουν τα αποτελέσματα της δημόσια διαβούλευση και ετοιμάζουν μια μελέτη αντικτύπου. Θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω για το ψήφισμά σα που σύστησε μια εναρμόνιση των ε, εργαλείων και μεθοδολογιών και ζήτησε να γίνουν υποχρεωτικές μελέτες αντικτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλω να προτείνω μια πρωτοβουλία πριν το τέλος του 2017 με σαφή ωφέλη για όλους και κυρίως ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφορά. τα 24 δίκτυα ε, που χρησιμοποιούν ε, λύσεις ε, ηλεκτρονικής ε, υγείας με συγκεκριμένο τρόπο. Παραδείγματο χάρη έχουμε συμβουλευτικά συμβούλια διασυνοριακά ε, για να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματά τους ασθενείς με σπάνιες ή σοβαρές αρρώστιες. Θα πρέπει αυτά τα δίκτυα να χρησιμοποιούν τηλεματικές υπηρεσίες ε, διασυνοριακά και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα ήθελα, θα ήθελα μαζί να προωθήσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το δίκτυο και να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του. Όπως ξέρετε, η ασφάλεια της υγείας και των τροφίμων είναι βασικό στοιχείο της ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινωνική συνοχή, η οικονομική ευημερία ε, συνδέονται με την υγεία. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική διάσταση της υγείας ε, στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο πυλώνας υιοθετήθηκε πέρυσι και προβλέπει ότι κάθε ένας έχει το δικαίωμα εγκαίρως να έχει πρόσβαση σε φθηνή περίθαλψη ε, και σε θεραπείες καλής ποιότητας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την πρόταση για μια διαθεσμική συνεργασία ε, για αυτό τον πυλώνα. Σας καλώ επίσης να συμβάλλετε επίσης στη συζήτηση για το, πάνω στο κείμενο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ανθρώπινη υγεία που είναι συμπεριφορά, περιβάλλον, κοινωνική κτλ. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες αρρώστιες και να μειώσουμε τους πρόορους θανάτους. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη σπατάλη των τροφίμων ως τμήμα των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως για τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις σπατάλες στα τρόφιμα και τις απόλυσεις θα πρέπει ε, να, ε, να γίνει μια προσπάθεια ε, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για αυτό το θέμα. Ελπίζω να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, κατευθύνοντας τις προσπάθειες ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ούτως ώστε να μειωθούν οι σπατάλες των τροφίμων μέχρι το 2030. Θα ήθελα τώρα να τελειώσω με ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Πιστεύω ότι το να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη το, τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ε, συνδέεται με τον εξυγχρονισμό του πλαισίου για την πολιτική μας για τα τρόφιμα και για ε, την εστίαση στο γενικό νομοθέτημα για τα τρόφιμα. Σήμερα, ε, με περηφάνεια, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το πιο πλήρες και αυστηρό σύστημα για διαχείριση των κινδύνων που αποτελούν τα τρόφιμα στο όλο τον κόσμο. Όμως η ποικιλομορφία των τροφίμων και η περιπλοκότητα των ε, διατροφικών, της αλυσίδας ε, ανεφοδιασμού σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια κρίσεις και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει μονίμως να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό έχουμε κάνει ε, ένα πλήρη έλεγχο καταλληλότητας για αυτό το γενικό νομοθέτημα για τα τρόφιμα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλο ακόμα. Θα μας βοηθήσει επίσης να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία αδυναμίας, ε, όπου θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και τα αποτελέσματα αυτής προσπάθειας θα δημοσιευθούν αργότερα μέσα στο 17. Ξέρω ότι έχετε πολλά ευαίσθητα θέματα ε, που σας απασχολούν. Δεν θέλω να μιλήσω για φυτοφάρμακα. Ξέρω ότι θα τα συζητήσουμε μέσω των ερωταποκρίσεων. Ξέρω θα μιλήσουμε για τους ενδοκρινικούς διαταράχτες και για όλα τα υπόλοιπα ευαίσθητα θέματα. Είμαι εδώ, είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Commission. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξή ε, Πρώτα οι συντονιστέ. και δύο λεπτά κάθε συντονιστή παρακαλώ ή δυνατόν να φύγετε δύο μόνο θέματα, όχι μέσα στην παρέμβασή σας να βάζετε πολλές, ε, πολλά στοιχεία, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο για τον Επίτροπο να σας απαντήσει. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε, μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά θα περάσουμε στον επόμενο γύρο των ε, ερωταπαντήσεων. Ε, Πρώτος ο κύριος Λίζη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε για αυτά που μας είπατε. Και ευχαριστούμε και για τη στράτευση που δείχνετε για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ λιγάκι θα ε, μιλήσω καθ' υπερβολή σήμερα. Γιατί αν δούμε λιγάκι ε, τις ε, προτάσεις, νομοθετικές προτάσεις ε, που υπάρχουν στην Επιτροπή μας και εμπίπτουν στις δικές σας τις ε, αρμοδιότητες. Παραδείγματο χάρη υπάρχει αυτή η έκθεση της κυρίας Γκρουστέτ για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στο Συμβούλιο και μίλησα με τον μελλοντικό πρόεδρο της Εστονικής Προεδρίας, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα ότι Όσον αφορά την Επιτροπή Γιούγκερ, μα η Επιτροπή αυτή ούτε, ένα προ, ούτε μία πρόταση δεν κατέθεσε. Ε, Βεβαίω και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην εκπονούμε πάρα πολλού κανονισμού, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειε, να μην επιβάλλουμε και υπαγορεύουμε στου ανθρώπου ε, τι επιτρέπεται να φάνε και τι επιτρέπεται να πιούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι νομοθετικέ πράξει. Φύγησαν δύο θέματα, αλλά θα ήθελα να σα παρακαλέσω να αγωνιστείτε έτσι ώστε εφέτος να έρθουν τουλάχιστον δύο συγκεκριμένες προτάσεις και όχι ε, προγράμματα δράσης. Στα αντιβιωτικά χρειαζόμαστε ένα εργαλείο, ε, χρειαζόμαστε να υπάρχει στοχευμένη δράση και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να δεχθούμε ότι χρειαζόμαστε και νέα αντιβιωτικά. Το Κοινοβούλιο σας έχει καλέσει επανειλημμένα να τοποθετηθείτε και αν δεν φταίτε ή αν δεν είστε εσείς αρμόδιος, επέστε μας ποιος είναι αρμόδιος για να έχουμε κάτι το συγκεκριμένο. Και το ίδιο ισχύει και για το Health Technology Assessment, HTA. Εδώ και τρία χρόνια μιλάμε για αυτό το θέμα και πρέπει να μας δώσετε μια συγκεκριμένη πρόταση. Όχι πρόγραμμα δράσης του τι θέλουμε να συζητήσουμε στο μέλλον, πρόταση. Δεν απευθύνομαι προσωπικά σε εσά, αλλά αν έχετε την καλοσύνη, πέστε μας με ποιο να συζητήσουμε για να γίνει και κάτι επί της ουσίας, κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόρτς, επόμενος ομιλητής. Ε, καλωσορίσατε, Επίτροπε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καταρχήν, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θα καταθέσει πρόταση σχετικά με τις ε, καλλιέργειες. Εγώ θα ήθελα να παραμείνω στα φυτοφάρμακα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη γλυφοσάτη. Γιατί υπάρχει μια θετική αξιολόγηση από την ΕΚΑ, αλλά υπάρχει και το έγγραφο της Μοντεσάντο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει με τη γλυφοσάτη. Και ε, τα ζυζένιοκτώνα. Ενδοκρινικοί διαταράκτες προφανώς και περιμένετε αυτή την ερώτηση από εμένα γιατί η συζήτηση στα κράτη-μέλη μέχρι τώρα δεν οδήγησε πουθενά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ε, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα που με ενδιαφέρει και φαντάζομαι το περιμένατε είναι ε, ο καρκίνος ε, πεπτικού συστήματος. Φαντάζομαι ότι θα περιμένετε να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το screening, για τη διάγνωση, όπως συνέβη και με άλλες οδηγίες Παραδείγματο χάρη για τον καρκίνο του μαστού, οι οποίες οδηγίες επικαιροποιήθηκαν. Ε, μιλάμε, όταν μιλάμε για τον καρκίνο του πεπτικού συστήματος, προφανώς μιλάμε και για τον καρκίνο του παγκρέατος, ε, που είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και θα ήθελα να γνωρίσω ε, πώς μπορούμε να έχουμε πρόληψη, θεραπεία του καρκίνου, του παγκρέατος, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να γνωρίζω αν ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να αντιμετωπιστεί ε, στο πλαίσιο των επόμενων οδηγιών που θα εκδώσετε για όλες τις μορφές ε, καρκίνου. Ίσως μπορείτε να θίξετε αυτό το θέμα και σχετικά και με τη χρηματοδότηση, γιατί μόνο το 2% ε, προβλέπεται για τη χρηματοδότηση έρευνας για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, ορισμένα θέματα και θα ήθελα ε, να αναφερθώ σε τρία εξ αυτών. Έχουμε λοιπόν μία έκθεση που αφορά ε, στα κτηνιατρικά φάρμακα και έγινε λόγος και για την ε, μικροβιακή εντοχή. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά δεν έκανε απολύτως τίποτα. αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, κτηνιατρικών φαρμάκων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει καλός συντονισμός. Σήμερα συζητήσαμε για την ε, επισήμανση των υνοπνευματοδών ποτών. Πρόκειται για ιδιαίτερα για ετικέτες, επισήμανση με μεγάλη εκκρίβεια, αλλά δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το ποια είναι ποιες είναι ενεργειακές τιμές ε, των υνοπνευματοδών ποτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολείται με αυτό. Παραδείγματο χάρη αναφέρεται η ε, περιεκτικότητα ζάχαρης, αλλά όχι άλλες ε, πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας και θέλει κανείς να διαβάζει στις, στις ετικέτες των προϊόντων. Και κάτι άλλο. Διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης το θέμα των ε, συμπληρωματικών ε, ουσιών ε, μιλάμε κυρίως για συμπληρώματα διατροφής. Από ό,τι φαίνεται, οι ουσίες αυτές υπάρχουν ε, και στα φάρμακα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λιγάκι το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Πράγματι, εγώ πιστεύω ότι ένα από τα θέματα που ετέθη είναι η γλυφοσάτη, το έγγραφο της Μονσάντος. Και η γλυφοσάτη είναι από τα πιο επικίνδυνα φυτοφάρμακα του κόσμου. Αυτό το έγραφο της Μονσάντο πώς ακριβώς επηρέασε τις μελέτες ε, τις οποίες ε, χρησιμοποιεί η ΕΦΣΑ, η ΕΚΑ αλλά και οι εθνικές αρχές επηρεάστηκε η άποψή του. Ε, κατά την άποψή του, η γλυφοσάτη προκαλεί καρκίνο, είναι καρκινογόνος ουσία, ναι ή όχι. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα φυτοφάρμακα, κυρίως ε, αυτά τα χαμηλού κινδύνου. Βλέπετε ότι στη Γεωργία γίνονται πάρα πολλές ε, κινήσεις ε, για να συμπεριληφθούν διάφορα φυτοφάρμακα, κυρίως αυτά τα χαμηλού κινδύνου. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, το ε, κατά πόσον ε, πράγματι στον γεωργικό τομέα μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας έστω αυτά τα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου. Και τρίτον, για να υπάρχει βιώσιμη ενεργεία, περισσότερο βιώσιμη λόγω της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας θρεπτικών ουσιών. Μήπως μπορείτε να βρείτε κάποιες εναλλακτικές λύσεις και για, την, για νέες μορφές καλλιεργιών. Η κυρία Κονιέτσινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θίξω μόνο ένα θέμα, το οποίο όμως είναι ύψης της σημασίας. Το 2015 σε αυτήν την Επιτροπή ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με την υπατήτηδα γάμα την φυματίωση και τον ιό HIV μέχρι το 2020. Στις 11 Απριλίου η Επιτροπή αυτή ενέκρινε μια δεύτερη προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή επί του θέματος. Και τι είδαμε, απολύτως τίποτα από τη δική σας πλευρά. Το μόνο που λάβαμε ήταν διαβεβαιώσεις, απλές ε, διαβεβαιώσεις. Ζητήσαμε διευκρινήσεις από τη Σλοβακική Προεδρία, τη Μαλτέζικη και η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται. Όλες οι στρατηγικές έχουν εκπνεύσει και στις όμορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν θετικοί φορείς ε, HIV και είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ασθένειες μέχρι το 2020 και για τη φυματίωση και για την υπατήτηδα γάμα. Όμως έγινε μία άτυπη συνάντηση στην Πρατισλάβα τον Οκτώβριο του 2016 και δεν έχει συμβεί τίποτα έκτοτε. Πότε θα αρχίσετε να κάνετε κάτι κύριε Επίτροπε, πότε θα προωθήσετε τα προγράμματα δράσης, πότε επιτέλους θα βοηθήσετε τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην υπεκφεύγετε συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Στάς. Ευχαριστώ Επίτροπε για την εισήγησή σας νωρίτερα. Έχει μεγάλη σημασία να τα λέμε για δεύτερη φορά ε, μέσα σε δύο-τρεις μέρες. Ακούσαμε, σας ακούσαμε και στο Βελγικό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη γλυφοσάτη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο η γλυφοσάτη και άλλα και άλλες πτυχές της πολιτικής σας. Η καταπολέμηση της χρήσης προϊόντων καπνού, η καταπολέμηση της παχυσαρκίας και ούτω καθεξής και ο συνάδελφος Μπότς ακριβώς γι' αυτό μίλησε. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ε, μόνο το γεγονός ότι είναι μία ε, καρκινογόνος ουσία, αλλά είναι και ένας ενδοκρινικός μεταλλάκτης, ε, πολύ επιζήμιος για τα ε, φυλαστικά και πλήττει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα γιατί ψηφίσαμε και στο Κοινοβούλιο πέρσι τον Απρίλιο και είπαμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, σε παιδότοπους και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπήρχαν τέσσερις όροι, τέσσερες συνθήκες. Ε, έπειτα η ΕΦΣΑ ε, βασίστηκε σε 182 μελέτες οι 82 δεν έχουν δημοσιοποιηθεί γιατί πρόκειται για εμπορικές πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα. Θα αλλάξετε επιτέλους τον κανονισμό για τα παρασιτοκτόνα, έτσι ώστε η ΕΦΣΑ να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή, αν οι βιομηχανίες μας δώσουν πληροφορίες, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί. Και εάν ορισμένες μελέτες δεν διατίθενται γιατί έχουν εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά, εν πρέπει να κινηθούμε στο δημόσιο τομέα με διαφάνεια. Νομίζω ότι έτσι εμείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και σε επίπεδο υπουργών. Η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τον Ιανουάριο του 2017 η σήμανση στη Γαλλία είναι υποχρεωτική τη στιγμή που υπάρχει περιεχόμενο κατά 50% ε, γαλακτοκομικών προϊόντων και 8% ε, προέλευσης κρέατος. Ξέρουμε ότι μας ε, επικρίνατε γι' αυτό και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει κάτι παρά, παρόμοιο για το βόλιο κρέας. Παρά τις επιφυλάξεις, δυστυχώς επεκτείνεται ο κατάλογος. Ο Ιταλός ε, ε, Υπουργός Γεωργίας μίλησε για παρόμοιες σημάσεις ως προς τα προϊόντα ρυζιού. Πώς προβλέπετε να επεκτείνεται αυτό το πλαίσιο σε σχέση με τη δράση των ΜΜΕ και ποια, ποιες ουσίες θα αποτελέσουν αντικείμενο παρόμοιων κανόνων. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ο πρώτος γύρος λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ξεκινάω με την ερώτηση του κ. Πίτερ Κλίζε για την μικροβιακή αντοχή και το σχέδιο δράσης, τα νέα αντιβιωτικά και τις συγκεκριμένες προτάσεις και την τεχνολογική τους αξιολόγηση. Όπως ανέφερα για την τεχνολογική αξιολόγηση, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης. Στη συνεχεία θα δρομολογήσουμε την μελέτη αντικτύπου και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε αφού σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Στο τέλος του 2017 ενδεχομένως θα κάνουμε και κάποια νομοθετική πρόταση. Εγώ είμαι υπέρ της μιας νομοθετικής πρότασης, αλλά πρώτα θα αξιολογήσουμε ολόκληρη την κατάσταση και θα δούμε αν θα κινηθούμε σε αυτή ε, την κατεύθυνση μετά τη μελέτη αντικτύπου. Για τη μικροβιακή αντοχή και τα νέα αντιβιωτικά, σήμερα υπάρχει μια πρωτοβουλία ε, για καινοτόμες μεθόδους και οι εταιρείε. Κάνουν κάποιες κλινικές δοκιμές. Υπάρχει πρόοδος σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης με κάποια πρώτα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε στην κοινή μας συνάντηση με τον Επίτροπο Υπεύθυνο ε, για τον τεχνολογικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, των κύριο Μουέδες. Τα μέτρα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο συνάδουν ε, με, το, την ουσία της πρότασής μας για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Ε, εσείς ζητάτε μια νομοθετική πρωτοβουλία. κοιτάξτε όμως τι γίνεται στα κτηνιατρικά φάρμακα. Πρώτα πρέπει να τελειώσουμε με τα κτηνιατρικά φάρμακα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, τελείωσε τα μαθήματά του, αλλά βλέπουμε το Συμβούλιο καθυστερεί. Θα πρέπει να σπρώξουμε το Συμβούλιο να είναι πιο ενεργό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, γιατί αυτά τα δύο μέτρα συνδέονται, αυτοί οι δύο τομείς συνδέονται. Και τον Ιούνιο θα προτείνουμε ένα νέο σχέδιο δράσης για να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή. Εγώ σας ζητώ ακόμα μια φορά να πιέσετε το Συμβούλιο για να είναι πιο δραστήριο στον τομέα αυτό. Τώρα, για την ερώτηση του κ. Πάβελ, για τα φυτοφάρμακα. Να ξεκινήσω με τα φυτοφάρμακα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολιτικός πώς. Όπως ξέρετε, έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές, email και τον Ιανουάριο υιοθετήσαμε την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου ε, υπογραφές, ούτως ώστε να απαγορεύσουμε τη γλυφοσάτη. Συμφωνούμε με την πρωτοβουλία. Είναι ένα καλό εργαλείο, ε, τουλάχιστον για να δημιουργήσει έτσι, και διαφάνεια και αφύπνιση στους πολίτες, περισσότερες συζητήσεις για τη χρήση γενικά των ε, φυτοφαρμάκων, όχι μόνο για το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο, τη γλυφοσάτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την παράταση της χρήσης της γλυφοσάτης για 7 χρόνια. Ε, εμείς με βάση την αρχή της προφύλαξης ζητάμε να αξιολογηθεί η κατάσταση για την καρκινογένεση της γλυφοσάτης. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα του φορέα ότι η γλυφωσάτη δεν είναι καρκινογόνο και δεν είναι μεταλλαξιογόνος ουσία, αλλά είναι τοξική για το αναπαραγωγικό σύστημα. Ξέρετε όμως ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αξιολογήσεις από την, ε, από, από την, ε, την οργάνωση του, του, του, του ΟΗΕ για τα τρόφιμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η γλυφοσάτη δεν είναι κακοινογόνα. Επίσης, ε, η, η, προστασία... η περιβαλλοντικής προφύλαξης της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας, της, ε, του Καναδά, από την ε, Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων της ε, Ιαπωνίας. Έχουμε πολλές επιστημονικές πληροφορίες. Έλαβα email από τις Ηνωμένε Πολιτείε, από τον Τζον Λίτλ, που είναι πολύ... από τη Ροσμαρή Μασόν, που είναι γνωστή ακτιβίστρια ε, ασχολείται πολύ με τα θέματα της Μονσάντο. Ε, στέλνει πολλές πληροφορίες. Εμείς τα στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες του στο Μοσάντο ε, για να υπάρχει διαφάνεια για αυτό το θέμα. Ε, Ξέρετε ότι το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι θέμα του χαρτοφυλακίου μου. και η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ ε, συμφωνούν ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί καρκινογόνα η γλυφοσάτη. Λαμβάνοντας αυτές τις επιστημονικές ε, γνώσεις υπόψη, ε, η γλυφοσάτη ε, πληρεί τα κριτήρια ε, όταν χρησιμοποιείται με προβλεπόμενο ρεαλιστικό τρόπο. Εμείς προτείνουμε ε, στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν, να υιοθετήσουν πιο αυστηρά πρότυπα για τη κλειφωσάτη. και πέρυσι συμφωνήσαμε σε επίπεδο επιτροπολογίας ότι θα πρέπει να τη μειώσουμε ε, τη γλυφοσάτη σε δημόσιους χώρους, στα πάρκα, τις παιδικές χαρές και να τη χρησιμοποιούμε όσο ε, να τον λιγότερο πριν από τη σοδιά. Επίσης προτείναμε να απαγορεύσουμε τη θαλιδομίδη, ε, που είναι επικίνδυνη μορφή. Επίσης ζητάμε, είναι επικίνδυνη ουσία. Επίσης ζητάμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το μηχανισμό βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων ε, και βιώσιμη διαχείριση των ζυζανίων. και να χρησιμοποιήσουν ας πούμε μη χημικές εναλλακτικές λύσεις όχι κατά ανάγκη φυτοφάρμακα. Αν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, ε, τότε θα μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τη χρήση τους. Ε, ορισμένοι με ρώτησαν για τα έγγραφα του Μονσάντο. Ξέρετε ότι ερευνάται η Μονσάντο στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Ξέρουμε ε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, το Dieselgate, ας πούμε, πολλά σκάνδαλα. Ε, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Αν αποδειχθεί όμως ότι αυτές οι μελέτες ε, πλαστογράφησαν επίτηδες στοιχεία, τότε θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, γιατί στην πραγματικότητα ε, παραβιάζονται όλες οι αρχές για καλές εργαστηριακές πρακτικές και αυτά είναι παραπίση στοιχείων κτλ. Και αυτό πρέπει να επισύρει νομικές συνέπειες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη, γιατί έχουμε νομική υποχρέωση να το κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα επιστημονικά στοιχεία και προτείνουμε στα κράτη-μέλη να συζητήσουν τα επόμενα βήματα έγκρισης, ίσως μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017. Ε, υπάρχει και η προσπάθεια ReFit γενικά για την νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα. Θα πρέπει να δώσουμε όλα τα στοιχεία για τα φυτοφάρμακα στα νομοθετήματα και αν χρειαστεί θα δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα νομοθετήματα για τα φυτοφάρμακα. Ίσως μέσω της διαφάνειας της ΕΦΣΑ, μέσω νέων δυνατοτήτων που θα απορρεύσουν από αυτή τη διαφάνεια. Θα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία πολύ προσεκτικά. Θα τα αξιολογήσουμε στο τέλος του 2017. για τα νέο νοικοτινοειδή χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα στα οποία έχει καταλήξει η ΕΦΣΑ. Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, γενικά για αυτά και για τα φυτοφάρμακα. Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες ε, Προστασίας των Τροφίμων αξιολογούν την κατάσταση και η προθεσμία ήταν ο Σεπτέμβριος του 2017 για τα νοικοτινοειδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν και είναι περίπλοκο το θέμα, πέρα από την αναθεώρηση. Όμως οι ετούντες ε, τους ζητήσαμε να δώσουν επιπλέον ε, στοιχεία για τα τρία νεονικοτινοειδή που επιτρέπονται ακόμα να χρησιμοποιούνται. Όλες αυτές οι, ε, οι τρεις ουσίες ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ περιορισμένους όρους και όσο επιτρέπει ο τρέχον κύκλος ζωής τους. Ε, αυτές τι τρεις ουσίες τι εξετάζει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Φυσικά η Κανονιστική Επιτροπή θα δώσει τη γνωμοδότησή τη για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, εγώ θέλω να τηρηθεί το δίκαιο, να ακολουθούμε μεγάλη αυστηρότητα τα επιστημονικά στοιχεία και να χρησιμοποιούμε την αρχή της προφύλαξης. Και θα παρακολουθούμε το σύνεγγι στην κατάσταση. Τώρα, για του ενδοκρινικού διαταράκτε, ήταν το ερώτημα, είναι το ίδιο θέμα ή συναφέ θέμα. Ξέρετε καταρχάς ότι γίνονται συζητήσεις με την ε, δική σα επιτροπή για τι προτάσει που θα κάνουμε για τα τελικά κριτήρια και τις ε, παρεκκλήσει. Και λάβαμε σαφεί απαντήσει από εσά ότι η Επιτροπή σας είναι υπέρ του διαχωρισμού των τελικών κριτηρίων και των από τις παρεκκλήσεις σε δύο διαφορετικά δηλαδή νομοθετήματα. Έτσι θα το κάνουμε. Αλλά δυστυχώς ε, έχουμε δύσκολε συζητήσει με τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ακόμα η ειδική πλειοψηφία για τα τελικά κριτήρια από τη μία. Και για τις παρεκκλήσεις από την άλλη επίσης δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Φυσικά ξέρουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο τα επιστημονικά στοιχεία, είναι και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Πρέπει να τα, τους δούμε και αυτούς. Μια και δεν έχουμε ειδική πλειοψηφία, δεν, υπάρχει, δεν έχει δώσει ε, γνώμη. Υπάρχει απουσία γνώμη στην ε, ε, Διαχειριστική Επιτροπή. Στην Επιτροπολογία δηλαδή. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε την ειδική πλειοψηφία. Ανησυχώ για την αρνητική αντίδραση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση ε, παρέκκλησης για τις επιλέξιμες ουσίες. Τώρα ε, σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματα και θα σας κρατούμε ενήμερους για το τι θα κάνουμε. Τώρα, για την έκθεση για την επισήμαση. Ε, το Μάρτιο υιοθετήσαμε μία έκθεση για την υποχρεωτική επισήμαση για τον κατάλογο συστατικών ε, στα αλκοολούχα ποτά. Ε, τώρα έχουμε... Δεν, δεν υπάρχουν λόγοι για να δικαιολογούν ε, παρεκκλήσεις υπέρ των αλκοολούχων ποτών. Να σας υπενθυμίσω το ότι η προηγούμενη πρόταση Κομισιόν ήταν η ίδια. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να δώσουν εξαιρέσεις ε, για τα αλκοολούχα ποτά. Σήμερα λοιπόν παρουσιάσουμε ακόμα μια φορά την έκθεση και λέμε σε αυτήν την έκθεση ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η παρέκκληση. Θα ζητήσουμε από τον κλάδι να παρουσιάσει τη δική του κοινή θέση. Ορισμένοι κατασκευαστές είναι υπέρ του να δίνουν την, ε, τις θερμίδες, το περιεχόμενο στην επισήμαση και άλλοι λένε όχι. Εμείς στην έκθεση λέμε όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινή στάση του κλάδου ε, και αν δεν είναι ικανοποιητική θα κάνουμε μια νομοθετική πρόταση. Για τα συμπληρώματα τροφίμων, ε, βιταμίνες και εχνοστοιχεία μέγιστα όρια ε, ε, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, ε, ενισχυμένα τρόφιμα κτλ. Ε, με βάση την νομοθεσία, το μέγιστο ποσό θα πρέπει να καθορίζεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις ε, τις επιστημονικές που κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων. Η χρήση ε, φυτών στα τρόφιμα και στα συμπλώματα τροφίμων θα πρέπει επίσης να ρυθμίζεται, αλλά σε εθνικό επίπεδο, με εθνικούς κανόνες απουσία ε, εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να κοινοποιούνται από την Κομισιόν. Αλλά βλέπω ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πολύ δραστήρια και θα ήθελα να υπάρξει συνεργασία και να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να κάνουν κάτι παραπάνω. Επίσης, ε, ε, για, τον, ε, για τον ιό του AIDS, εγώ απάντησα για τη φυματίωση. Έχουμε πάρα πολλούς ε, συναντήσεις. Εγώ συναντήθηκα με αρμόδιους στις χώρες. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών. Ξέρετε ότι τα βασικά προβλήματα υγείας είναι θέμα των κρατών μελών. Θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να καταπολεμήσουν τις πιο χοντρές ε, ανισότητες. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες για να προωθηθούν ε, εθνικά προγράμματα υγείας, για να δοθούν απαντήσεις ε, για ευάλωτες ομάδες. Ε, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για την, για την ναρκωτικά και την τοξικομανία που έχει εντοπίσει καλές πρακτικές και κενά και παρεμβάσει πρέπει να γίνουν. Προσπαθούμε να διαδώσουμε αυτές τις πρακτικές, ούτω ώστε να δώσουμε πληροφορίες στα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που υπάρχουν. Θα προωθήσουμε ε, την ε, ανανέωση ενός think tank που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ιό του για να σκέφτεται πρακτικές, καλύτερες πρακτικές ε, και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποιες ασυμμετρίες ανάμεσα στη συνθήκη της Λισαβόνας Έχουμε τα μέτρα για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, το συντονισμό, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν παραπάνω πράγματα για να έχουμε κοινέ δράσει και χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Εγώ με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τη δική σα τη συνεισφορά, να πιέσετε κι εσεί τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν και να εξτάσουν αυτά τα θέματα. Υπάρχει και το θέμα την, ε, της επισήμανσης ε, σχετικά με την πρόελευση. Εμείς ε, περιμένουμε τη γαλλική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της επισήμανσης μέχρι τα τέλη του 2018. Και μετά θα αξιολογήσουμε το επόμενο βήμα μας, γιατί χωρίς να έχουμε στα χέρια μας κάποια ανάλυση δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ε, θα πρέπει να μιλήσετε κατά το μέγιστο ένα λεπτό. Πάρα πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο και πρώτος ομιλητής ε, στον κατάλογό μου είναι η κυρία Γκρουστέτ. Λυπάμαι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθούμε και στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Έχουμε ένα συμβούλιο που παραλύει τα πάντα. Ε, συζητάει επί μακρόν τη στιγμή που έχουμε ε, να κάνουμε με κατεπήγοντα θέματα, όπως την ε, μικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει τα πράγματα πιο γρήγορα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, εναρμόνωση της νομοθεσίας για τις ιατρικές τεχνολογίες. Θα μας υποβάλλετε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με τα παιδιατρικά φάρμακα θα θέλαμε τα αποτελέσματα της μελέτης σας, τα περιμέναμε για την Άνοιξη, τώρα θα τα έχουμε μετά το καλοκαίρι. Και ως προς τους παιδικούς και εφηβικούς καρκίνους θα πρέπει να τύχουν ειδική μεταχείρισης. Θα πρέπει να προβάλλουμε ένα πρόγραμμα δράσης μόνο για τους παιδικούς και εφηβικούς καρκίνους όπως ίσχυε στο παρελθόν για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ. Ο κύριος Παρνιό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων που βρίσκεται στο Λονδίνο θα πρέπει να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν από, την, ε, από το Συμβούλιο της 29ης Απριλίου είπαμε ότι, είδαμε μάλλον ότι δεν ελήφθη απόφαση ακόμα. Μπορείτε να μας πείτε τι υπόθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο για την μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Μπορείτε επίσης να μας πείτε κατά πόσο το Συμβούλιο αναφέρθηκε στα κριτήρια αξιολόγησης γιατί μπορεί να ζητηθεί η γνώμη και της Κομισιόν για τις υποψήφιες χώρες. Στις 19 Απριλίου η γαλλική κυβέρνηση πρόβαλε την πόλη της Λίλης ως υποψήφια για τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και εγώ υποστηρίζω αυτή την υποψηφιότητα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι η Λίλη βρίσκεται κοντά στο Λονδίνο, μία ώρα και είκοσι είναι η, η ώρα για τη μετάβαση από τη μία πόλη στην άλλη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η υποψηφιότητα έχει μεγάλη σημασία και για τους 900 ε, μισθωτούς που θα βρίσκονται κοντά στο Λονδίνο. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Χαίρετε. Στις 11 Ιανουαρίου έγινε μια παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με μια έκθεση για το ε, JRC. Και ε, τα συμπεράσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ε, δεν υπάρχουν ε, θετικές επιδράσεις από την απαγόρευση των νέων νοικοτινοειδών. Δηλαδή δεν ε, ευημερεί η μέλισσα μετά την απαγόρευση ή οποιαδήποτε άλλα έντομα. Και αυτό σχετίζεται και με την κατάσταση πριν από την απαγόρευση σε ένα ή δύο κράτη-μέλη που είχαν προαπαγορεύσει τα νεονικοτινοειδή και είδανε ότι υπήρχε, υπήρχαν οι ίδιες επιπτώσεις στην υγεία των επικονιαστών. Εγώ έχω το PowerPoint αν θέλετε, αλλά δεν μας δόθηκε η έκθεση, η οποία φαίνεται τώρα ότι δεν είναι διαθέσιμη, δεν τη λάβαμε από το JRC, ούτε από την ΕΦΣΑ. Και θα ήθελα τουλάχιστον να τη λάβω από εσάς, γιατί έχει δημοσιευθεί αλλά έχει αποσυρθεί. Αν και είπατε ε, τώρα προβάλλεται μία νέα απαγόρευση για τα ε, νεονικοτινοειδή και δεν φαίνεται ότι οι τρεις ουσίες ήταν ήδη επιτυχείς. κυρία Βιέντνικ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, θα ήθελα υποβάλω μία ε, ερώτηση από πλευράς της κυρίας Μάισνερ θα ήθελε και Μάισνερ να ασχοληθούμε με αυτό το ε, θέμα και μετά τις διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή εφαρμογή των κανονισμών για τα φάρμακα. Έχει μεγάλη, έχουν μεγάλη σημασία οι πόροι καθώς και η κατεξουσιοδότηση πράξης. Ορισμένες κατεξουσιοδότηση πράξεις είναι προαπαιτούμενο πριν από την εφαρμογή του κανονισμού για τον ιατρικό εξοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε πώς η διαδικασία κοινοποίησης θα ολοκληρωθεί. Επειδή η μεταβατική περίοδος είναι τριετής, η οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση θα οδηγούσε σε καθυστέρηση προσαρμογής από του, τους κατασκευαστές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς, έχουν αυτές, πώς έχει αυτός ο εξοπλισμός στην αγορά, ο ιατρικός εξοπλισμός και πώς η Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή για να μην υπάρξουν ελλείψεις και να μπορούμε να παρέχουμε τη θεραπεία στους ο κύριος Μπέκ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έγκριση της έκθεσης πρωτεβουλίας μου για τις ελάχιστες προτρεχές σχετικά με την εκτροφή των ε, ε, κουνελιών ότι στην εκτροφή των κουνελιών χορηγούνται μαζικά αντιβιωτικά. Γιατί τα κουνέλια είναι ευεπίφορα, είναι επιρρεπή στο να δεχτούν ασθένειες. Προσβάλλονται πολύ εύκολα από ασθένειες. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την εκτροφή σε κλοβούς και με τα αντιβιωτικά μπορούν να περιστούν κάποιες ασθένειες. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε σας ερωτώ κατά πόσον συμφωνείτε με αυτά που είπε η συνάδελφό σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, κύριο Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, αυτές οι χώρες που εκτρέφουν κουνέλια, αυτές να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, πιστεύετε κι εσείς ε, ότι η μικροβιακή αντοχή η οποία μπορεί να ξεκινήσει από την εκτροφή των κουνελιών. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο ή θα ήταν καλύτερα να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ριβάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας, γιατί έχουμε πολλές ανησυχίες ε, Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 17 και το 2014 είχαμε πάντα το πρόβλημα των ε, ενδοκρινικών διαταρακτών και δεν έχουμε καμία πρόοδο. Δεν έχετε την ειδική πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και οι προτάσεις επιτροπής που μπλοκάρουν το σύστημα. Ως προς τη γλυφοσάτη, εδώ θα ήθελα να προχωρήσουμε και έχετε σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη γνωμοδότηση ενός οργανισμού εάν δεν υπάρχει open access σε όλες τις μελέτες. Γιατί στη νέα οδηγία για το copyright υπάρχει open access. Και εδώ θα πρέπει να πείτε στην ΕΦΣΑ ότι εάν δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις μελέτες δεν θα τις λάβουμε υπόψη. Ε, έτσι πολυεθνικές θα αναγκαστούν να τις δημοσιεύσουν. Επίσης, ως προς τα ε, νανομόρια στις ε, τροφές, πώς, βρέθηκαν, ε, πώς βρέθηκε διοξίδιο τιτανίου στις τσίχλες, στις καραμέλες και στο λευκό κρέας, ενώ ο κανονισμός 1069 ε, επιβάλλει την επισήμανση. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να παρέμβει σε επίπεδο κρατών μελών για να είναι υποχρεωτική η σήμανση. Πώς μπορούμε να έχουμε διοξίδιο του τιτανίου στις καραμέλες και να μην ε, ε επισημαίνεται. Στη Γαλλία αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα των ταμπών, των γυναικείων ταμπών, όπου υπάρχουν διοξίνη και παρασιτοκτόνα και μας λένε ότι οι βιομηχανίες δεν αναγράφουν τα συστατικά στοιχεία. Θα ήθελα να μάθω γιατί. Εάν έχετε άλλα ε, θέματα, να τα δείξετε στην Ολομέλεια. Τώρα όμως πρέπει να σταθούμε στο ένα λεπτό. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Ε, θα έλεγα να χρησιμοποιούμε όλοι τις λέξεις με την ίδια έννοια. Άκουσα ότι να χρησιμοποιείται ο όρος ε, φυτοφάρμακα και μάλιστα και από τον κύριο Επίτροπο. Αλλά εδώ πρόκειται για ζυζανιοκτώνα. Ε, πολλές φορές μιλάμε και τα μπερδεύουμε. Άλλο ζυζανιοκτώνα, άλλα παρασιτοκτώνα και εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά θέλω να είμαι και ε, πολύ προσεκτική. Η γλυφοσάτη λοιπόν σκοτώνει τα παράσιτα. Ε, με ενδιαφέρει η κοινή γνώμη και όσον αφορά την ε, δική μου τη γνώμη, και εγώ γνώμη για πολλά θέματα, αλλά δεν έχω πολλές φορές τεκμηριωμένη γνώμη. Εσείς ε, τι μπορείτε να πείτε στους επιστήμονες ε, οι οποίοι αναλύουν τις μελέτες. Ελπίζω αυτό να σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί η κοινή γνώμη μπορεί να είναι παραπλανητική. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η ειδική τεχνογνωσία. Τώρα, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σημαντικός, σημαντική έδρα του, αλλά το πιο σημαντικό μετά το Brexit είναι ο οργανισμός αυτός να συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των πολιτών. Ε, ξέρω ότι αναφέρθηκε η Λίλη, αλλά και γιατί όχι το Δουβλίνο. Μια χαρά είναι το Δουβλίνο. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ. Κυρία Μπόρζαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Εγώ είμαι το σημείο επαφή Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με, τη, με την κατάστασή του, όπως ρώτησε ήδη ο Συνάδελφο μου Ζιλ. Ερώτησε για το μέλλον αυτού του οργανισμού, ε, για τι συζητήσει που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο σε επίπεδο ε, κορυφής. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το κτίριο. Και αυτό θα ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Brexit. Ξέρουμε επίσης ότι ο οργανισμός αυτός θα χρειαστεί επιπρόσθετα κονδύλια για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του ε, χωρίς καμία αναστολή. Προβλέπετε λοιπόν ε, να ε, υπάρξει έξτρα χρηματοδότηση αυτού του οργανισμού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ έχω μια τελείως ε, διαφορετική ερώτηση. Τεχνικά, τεχνικά ε, λιβάδια. Τεχνητά λιβάδια, με συγχωρείτε. Έχει μια μελέτη σχετική. Ε, τεχνητά λιβάδια υπάρχουν και μας ε, στη Φλάνδρα με SPR κόκκους, κόκκι που προέρχονται από χρησιμοποιημένα ελαστικά. Και αυτοί οι κόκκι είναι καρκινογόνοι. Η Κομισιόν λέει, υπάρχει μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Ουσιών, ΕΚΑ, και η μελέτη καταλήγει ότι θα πρέπει να περιοριστεί αυτή η χρήση αυτών των κόκκων. Αλλά η άποψη είναι ότι ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ΕΚΑ όμως λέει στην ε, Κομισιόν να τηρούνται οι προδιαγραφές του κανονισμού REACH. Εγώ ερωτώ, μήπως θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τις ε, προδιαγραφές του κανονισμού REACH. Εσείς ποια είναι η αποψή σας σχετικά με αυτές τις τελευταίες πληροφορίε που προέκυψαν από την ΕΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Κύριε Πίτροπε, εγώ θα διαμαρτυρηθώ για την ολιγορία και απραξία τη δική σα και της γενική σας διεύθυνση, διότι εγώ σας είχα στείλει μια επιστολή να μας πείτε τι είναι τα φυτικά τρόφιμα, γιατί αυτό το χρειαζόμαστε ε, και μας ε, πήρατε, μας είπατε έχουμε άλλες δουλειές τώρα, έχουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες, ε, θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα και είπατε ας πούμε για μία διορία για ένα πράγμα όμως το οποίο είχε εκπνεύσει πριν από δύο χρόνια όπως είχε εκπνεύσει και για τα υνοπνευματώδη ποτά. Κατόπιν τούτου, η πρόταση για τα υνοπνευματόδη ποτά, ξέρετε, εγώ είμαι σαφώς υπέρ της ε, ανάληψης ευθυνών, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς ε, μικρές επιχειρήσεις ε, στον τομέα των πνευματοδών θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με το ότι ένας ολόκληρος ε, τομέας μέσα σε ένα χρόνο αναλαμβάνει μόνο στο να ρυθμίσει τα θέματα της θρεπτικής αξίας. Επίσης, ο ορισμός των μερίδων είναι πολύ σημαντικό γιατί το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτός ο ορισμός που πρέπει να γίνει από την Επιτροπή αυτό έχει οδηγήσει στο ότι με πέντε μεγάλοι όμιλοι τροφίμων έχουν σκεφτεί ένα δικό του σύστημα επισήμανσης ένα σύστημα που βασίζεται σε μερίδες τα οποία αυτοί τα ορίζουν μόνοι τους και αυτό είναι πάλι παραπλανητικό για τον καταναλωτή Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα πρέπει κάτι να κάνετε, επιγόντως απαραίτητο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τελευταίο θέμα, το θέμα της ετικετοθεσίας και της ε, διατροφικής ασφάλειας. Νομίζω ότι δεν ασχοληθήκατε παρκώς με το θέμα αυτό. Ε, όπως και με το θέμα της, α, ε, μερικές φορές αυτή η ισχυρισμή πούμε, για τη διατροφική σημασία είναι παραπλανητική διαφαίνηση. Εγώ θα ήθελα να μιλάτε για διατροφικό προφίλ και μετά να με βάση το οποίο θα μπορεί να επιλέγει ο καταναλωτής. Επίσης, το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με απασχολεί. Ε, μελετάμε την επίπτωση που θα έχει η όποια αλλαγή. Ε, είναι σημαντικό να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία σωστά. Επίσης, ε, το σχέδιο για τη μικροβιακή αντίσταση θα, θα εκδοθεί τον Ιούνιο. Ε, δεν κατάλαβα καλά από την παρέμβαση της Κομισιόν. So, thank you very... Ευχαριστώ. Κλείνει ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ο Επίτροπος. Έχω λάβει ένα κατάλογο. Αλλά δεν έχουμε ε, δεν έχουμε χρόνο για να δώσω το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο για όλα αυτά ονόματα στον κατάλογο. Απλώς δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη. Μπορεί να σας στον κατάλογο, αλλά ο κατάλογος ήταν πάρα πολύ μακροσκελής. Εγώ το εξήγησα στη συνάδελφο, λυπάμαι που δεν σα το είπε και σας έγραψε παρόλα αυτά στον κατάλογο. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από την ερώτηση της κυρίας Γκοστέτα. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι πολύ απογοητευτική η κατάσταση. Απογοητευτικότατη ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Το θέμα όμως είναι πολύ τεχνικό, αλλά όχι μόνο τεχνικό. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για όλα τα θέματα, με, θα δουλέψουμε με διαφανή τρόπο. Ξέρετε ότι μερικές φορές ε, για να πάρει κανείς κτηνιατρικά φάρμακα χρειάζεται συνταγή. Και για να πουλήσει κτηνιατρικά φάρμακα και για να αγοράσει κτηνιατρικά φάρμακα χρειάζονται άδειε. Ε, Φυσικά είναι δύσκολο να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να μειώσει τη χρήση των ε, κτηνιατρικών φαρμάκων. Για την αξιολόγηση ε, της για την υγεία. Ε, καταρχάς έχουμε κάποιες πρώτες, ε, κάποια πρώτα... Η πρώτη αξιολόγηση μετά τα σχόλια που λάβαμε από τη δημόσια διόλευση είναι πολύ ενθαρρυντική. Οι περισσότεροι stakeholders θέλουν ενισχυμένη συνεργασία για την αξιολόγηση αυτή του, της τεχνολογίας για την υγεία και μετά το 2020. Ξέρω βεβαίως ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ διάφορες χώρες και να συζητήσω με υπουργούς για την προσέγγιση τους. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε τη μελέτη αντικτύπου και μετά θα δούμε ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο συνολικά. Γιατί πρέπει να έχουμε ευρύτατη συνένεση. Αλλά η δημόσια διαβούλευση έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επίσης, χαίρομαι για το ενδιαφέρον σα ε, για το θέμα των φαρμάκων για τα παιδιά. Ε, εμείς ετοιμάζουμε μία δεύτερη έκθεση για τον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα. Έχουμε λάβει κάποια δεδομένα το Φεβρουάριο του 2017 και τώρα θα πρέπει να τα αναλύσουμε και θα ετοιμάσουμε την έκθεση μέχρι το τέλος του 2017 ε, πριν Επίσης θα ετοιμάσουμε και μια περίληψη με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Όλα αυτά θα είναι δημόσια, δημοσιοποιημένα γιατί θέλουμε καλή συνεργασία και διαφάνεια. Ξέχασα να απαντήσω στον Πάβελ για τον παγκρεατικό καρκίνο, για τον καρκίνο του παγκρέατος. Θα σταθώ χωριστά σε αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε με πολλές λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό και λεπτομερές. Και μια άλλη ερώτηση από τον κύριο Παγνιού. Ξέρετε ότι η Κομισιόν εκπονεί αντικειμενικά κριτήρια. Όλα τα τεχνικά στοιχεία τα λαμβάνει υπόψη. Και ο κύριος Γιούνκερ ε, συζητάει αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο Ντόναλτ Τούσκ για να αποφασίσουν ε, αν θα συζητήσουν αυτά τα θέματα ενδελεχώς τον Ιούνιο στο Συμβούλιο στον Ιούνιο θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Μην με ρωτάτε τώρα για ποιες πόλεις, για ποιες χώρες. Δεν απόκειται σε εμά. Είναι στα χέρια του Συμβουλίου το θέμα. Εφτά με έντεκα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται τα μεν τα δε. Το καταλαβαίνω. Καταρχάς πρέπει να έχουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις ε, υποχρεώσεις μας. Για να προστατεύσουμε την υγεία των ασθενών, να εξασφαλίσουμε μία συνέχεια και να υπολογίσει όλες τις συνέπειες στο Συμβούλιο. Ε, όχι μόνο τις οικονομικές συνέπειες. Φυσικά και τα οικονομικά το Συμβούλιο αποφασίζει. Το ξέρουμε πολύ καλά και μόνο αφού ληφθεί απόφαση θα δούμε όλα τα τεχνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα κτλ. Και θα μας παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα, το Συμβούλιο δηλαδή. Η Κομισιόν είναι ουδέτερη στο θέμα αυτό. Τώρα, για τον Οργανισμό Φαρμάκων. Θα απαντήσω συνολικά. Κοιτάξτε, το θέμα δεν έχει καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Είναι εσωτερικό θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Ένα άλλο ερώτημα. Για μια έκθεση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Πήγα την περασμένη εβδομάδα στη Σεβίλη και είχα την ευκαιρία να συζητήσω αυτά τα θέματα. Σας ευχηστώ την προσοχή στο εξή ότι αυτή η μελέτη δεν έγινε γιατί υπάρχει αντίρρηση με τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ. Γίνονται συζητήσεις για τις διαφορετικές ε, δυνατότητες που έχουμε στο μέλλον τα οικονομικά θέματα, τη συμπεριφορά των αγροτών και θα ζητήσω το, από τον Τζέρσι να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, ε, η έκθεση αυτή δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν έχουν γίνει οι επιστημονικές μελέτες για τις μέλισσες και την ε, αλλαγή πρακτικών ως προς την, ε, τις ουσίες που χρησιμοποιούνται από τους ε, ε, γεωργούς. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφή και εγώ θα ακολουθήσω την επιστήμη και θα προστατεύσω τις μέλισσες, γιατί καθίσταται απόλυτα σαφές ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν εις βάθος. Να δούμε δηλαδή πώς θα αντικαταστήσουμε τα ζυζανιοκτώνα με τα παρασιτοκτώνα. Ποια είναι πιο τοξικά κατά των μελισσών. Έγινε λόγος και για την προστασία των κουνελιών. όλα τα είδη προστατεύονται από την Οδηγία 98 κάθετος 58, έτσι ώστε να μην υφίστανται ε, πόνο όλα τα ζώα. Και επειδή για τα κουνέλια δεν υφίσταται μια τέτοια διαδικασία, δεν έχουμε προβάλει ένα συνολικό μέτρο. Όμως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των κουνελιών μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, πλατφόρμας και να γίνουν έλεγχοι και να δούμε πώς έχει η κατάσταση επιτόπια σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις και θα ζητήσουμε από τις ε, υπηρεσίες μας να γνωμοδοτήσουν μετά από τον έλεγχο. Αλλά η πλατφόρμα της ευημερίας των ζώων είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα συζήτησης και θα ζητήσουμε την υποστήριξη των κρατών μελών επί του θέματος. Η κυρία Βέρνικα μίλησε για τον ιατρικό εξοπλισμό. Όπως ξέρετε, η Επίτροπος Μπενκόφσκα είναι υπεύθυνη επί του θέματος. Όπως είπα τον Απρίλιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, εγκριθεί η οδηγία για τον διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισμό. Και τα δύο αυτά κείμενα αποτελούν την απαρχή μιας ε, μακράς διαδικασίας. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τους ασθενείς, τους ιατρούς, ε, τους οργανισμούς και τον ε, ιατρικό ε, εξοπλισμό θα τύχουν σύγκλησης και η κυρία Μπιενκόφσκα καθώς και οι δικές μου υπηρεσίες θα δώσουν ένα follow-up τη διαδικασία σε σχέση με τα νανοσωματίδια ε, προσπαθούμε να εργαστούμε με βάση τις κατεξουσιοδότηση πράξεις για τους καταναλωτές. Ο κύριος Ζόμπερς μίλησε για το refit και την διατροφική αξία των τροφίμων μέσα στα πλαίσια της ε, χρηστής ε, ρύθμισης και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε ε, υπόψη ε, την θρεπτική αξία των, ε, των ουσιών και αυτό εν ώψη του 2018. Δεν είναι σκόπιμο να φτάσουμε σε συμπεράσματα τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Βεβαίως οι χορτοφάγοι ανησυχούν ιδιαίτερα, όμως θα προβούμε σε αυτή την αξιολόγηση σε σχέση με τη θρεπτική αξία των ουσιών. Ο κύριος Μάκερ μίλησε για το, για το το οποίο ε, ε, έχει μεγάλη σημασία και μέσα στα πλαίσια της εντολής που έχουμε. γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω μια τέτοια ερώτηση. Νομίζω ότι συνόψισα. Α, συμφορώ με την κυρία ε, Μαγκίνες. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε για παρασίτοκτόνα να μιλάμε για ζυζανιοκτώνα, φυτοκτώνα και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το γενικό όρο παρασίτοκτόνα, διότι ενέχουν διαφορετικές χημικές ουσίες, γιατί ε, μιλάμε για παρασίτοκτόνα γενικά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η στοχοθέτηση. Υπάρχει μεγάλη ρήξη μεταξύ επιστήμης και ανθρώπων. Ο Γαλιλαίος μας είχε πει ότι η γη κινείται, κινείται γύρω από τον ήλιο, αλλά τότε η κοινή γνώμη δεν ήταν υπέρ και ο Κοπέρνικος έκανε το ίδιο, γιατί ξέρουμε ότι η κοινή γνώμη ήταν πολύ επικίνδυνη τότε. Τώρα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε τους επιστήμονες να είναι ανοιχτοί και να εκφράζονται και να συνομιλούν με την κοινωνία γιατί δυστυχώς ε, αν ε, είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την επιστήμη τότε δεν μπορούμε να προωθήσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας γιατί μιλάμε για τον εμβολιασμό, για παράδειγμα. Και εκεί υπάρχει το θέμα της κοινή γνώμης. Πολλοί είπαν ότι ε, τα εμβόλια και ο εμβολιασμός προκαλούν τον ε, αυτισμό και αυτό οδήγησε σε λανθασμένα αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για τη γλυφοσάτη. Αυτές οι μελέτες δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένες, χρειάζεται μία δημόσια συζήτηση. Μιλάμε για νέες τεχνικές και θα γίνει μια μεγάλη διάσκεψη το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες όπου θα καλέσουμε τους πάντες για να μιλήσουμε για θέματα νέων τεχνικών καλλιέργειας. Γιατί τώρα έχουμε δημοσιεύσει την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για τις νέες καλλιέργειες και θα πρέπει να διαβάσετε αυτή την έκθεση για να δείτε πώς προοδεύει η επιστήμη. σε σχέση με 20 χρόνια πριν πολύ διαφορετική κατάσταση σήμερα σε σχέση με τους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Θα πρέπει να συζητούνται αυτά τα ζητήματα. Εγώ είμαι συνήγορος της επιστήμης. Της επιστήμης. Δεν μπορώ να μην με την επιστήμη.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 η εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με, τον, με την ενημέρωση. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός ή αν θέλετε υπάρχει ε, πολύ μεγάλη καθυστέρηση ακόμα και αν στον κανονισμό υπάρχουν προθεσμίες και με τη δικαιολογία ότι καταρχήν θα πρέπει να επεξεργαστούμε όπου, έχουν υπάρξει, όπου υπάρχουν προθεσμίες. Ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν προθεσμίες το χρησιμοποιείτε σαν δικαιολογία και δεν κάνετε τίποτα άλλο. Αυτή λοιπόν η καθυστέρηση οδηγεί οδηγεί σε νομική ασάφεια και όχι μόνο αυτό, αλλά το μεταξύ και σε παραπλάνηση του καταναλωτή. σα την ερώτηση. Νομίζω ότι με ρωτήσατε για τις ε, εκτελεστικές πράξεις που συνδέονται με αυτόν τον κανονισμό. Σωστό? Ναι. Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις, ε? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα το τσεκάρω, θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω. Γιατί θέλω να δω σε τι φάση είμαστε. Ξέρω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι και μια δουλειά πολύ χρονοβόρα. Λυπάμαι που σας το λέω έτσι, αλλά πραγματικά δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω. Δεν σας κατάλαβα καλά για τις εκτελεστικές πράξεις μας, ε, με ρωτούσατε. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, που ήρθατε. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, που συμμετείχατε στη συζήτηση. Σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε.